Uh, good afternoon everybody and uh, Καλώς ορίσατε στην ακρόαση που οργανώνουμε σήμερα το απόγευμα. Μπορείτε να καθίσετε. Έχουμε πολλές κενές θέσεις. Καθίστε, καλώς ορίζω όλους τους ε, επισκέπτες. Πρέπει να ξέρετε ότι γίνεται αναμετάδοση της σημερινής ακρόασης και θέλουμε όλοι όσοι ενδιαφέρονται να μπορέσουν να υποφεληθούν. Έχουμε πολλά μέλη της κοινότητας των μοτοσυκλετιστών που προσβλέπουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην συζήτηση που έχουμε σήμερα εδώ, έτσι ώστε να εξετάσουμε τα θέματα αυτά. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι υπάρχει και μία ιστοσελίδα και μία διεύθυνση ηλεκτρονική, αν θέλετε να μας ε, στείλετε σχόλια ή παρατηρήσεις ιδιαίτερα προς τον εισηγητή μας, ο οποίος συνεχίζει να εργάζεται το θέμα αυτό, βρίσκεται δίπλα μου. Επίσης υπάρχει και ο σύνδεσμος για να έχετε επαφή με μας και με την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Είμαι σίγουρος ότι μετά από αυτή την ακρόαση θα θελήσετε να γίνετε φίλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς. Έχουμε τις σημερινές παρουσιάσεις, μπορείτε να τις πάρετε. Έχουμε το σημερινό πρόγραμμα. Θα σας παρουσιάσω τους ομιλητές όπως προχωράει η ακρόαση. Σκοπός μας είναι σήμερα να συζητήσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση των, του κανονισμού όσον αφορά την εποπτεία και την εσωτερική αγορά για τα δίκυκλα, τρίκυκλα και τις μοτοσικλέτες. Είμαστε, όπως ξέρετε, αρμόδιοι από κοινού τις 27 κυβερνήσεις, οι οποίες επίσης εξετάζουν αυτήν την πρόταση κανονισμού. Είναι εδώ βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλωσορίζω τον κύριο Ζων Φιλιππιό, που είναι εδώ επικεφαλής της αρμόδιας διεύθυνσης της ε, Επιτροπής. Ε, σας καλωσορίζω και εσάς και τους συνεργάτες σας. Ο εισηγητής, ο οποίος έχει οριστεί από την Επιτροπή μας, υπεύθυνο για το θέμα αυτό, κάθεται αριστερά μου. Είναι ο κύριος Βίμαν Τεκάμπ, ο οποίος θα πάρει το λόγο λίγο αργότερα και θα μιλήσει για την πρότασή του. Θέλουμε σήμερα να ακούσουμε ειδικού, να ακούσουμε προτάσεις για τα θέματα που μας αφορούν. Η Επιτροπή έχει εξετάσει το υπάρχον καθεστώς και είναι σήμερα προφανές ότι χρειάζεται αναθεώρηση για θέματα που αφορούν την ασφάλεια, το περιβάλλον, τις περιβαλλοντολογικές επιδόσεις για αυτή την κατηγορία οχημάτων και βεβαίως θα γίνει και μια συζήτηση για το χρονοδιάγραμμα και για την ε, ικανότητα του κλάδου των ε, δικύκλων, των μοτοσυκλετών όσον αφορά τις επισκευές, τα ανταλλακτικά. Υπάρχουν δηλαδή και σοβαρά οικονομικά θέματα. Αυτά είναι τα εισαγωγικά μου σχόλια. Έχουμε στη διάθεσή μας δύο ώρες μέχρι τις 6.30. Θα ήθελα να ζητήσω καταρχήν από τον εισηγητή, ο οποίος εργάζεται σκληρά, να μας παρουσιάσει το θέμα. Με μεγάλη χαρά σας δίνω το λόγο, κύριε Σεγητά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να σας πω ότι έχω προετοιμάσει μια μικρή παρουσίαση για σήμερα το απόγευμα με έναν πολύ ωραίο τίτλο. Έχετε την παρουσίασή μου στους φακέλους σας. Βεβαίως, θα κάνω κάποια εισαγωγικά σχόλια. Καταρχήν, νομίζω ότι όλοι γνωρίζετε το χρονοδιάγραμμα Πρέπει να σας πω ότι αναγκάστηκα να το τροποποιήσω. Η διαδικασία αυτή έχει άμεση σχέση με τον κανονισμό ο οποίος εφαρμόζεται για τα μηχανήματα στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομείας. Υπάρχουν λοιπόν σήμερα πολύ σημαντικές καθυστερήσεις γιατί το Συμβούλιο έχει εκφράσει την επιθυμία του να υπάρξει ο ίδιος ρυθμός για τα γεωργικά μηχανήματα, για τα μηχανήματα που αφορούν την δασοκομεία, αλλά και τις μοτοσυκλέτες, τα σκούτερ, τα μοτοπολίδηλατα. Βλέπετε λοιπόν εδώ το χρονοδιάγραμμα όπως έχει παρουσιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα, θα το ονομάσω προκλήσεις, που αφορούν πάντα τα μηχανήματα, τα γεωργικά και θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας όσον αφορά τις διάφορες μεθόδους εργασίας, τις εκπομπές γύρω 5, γύρω 6, γύρω 7, το OBD, διάγνωση επί των οχημάτων, κάτι το οποίο φαίνεται εδώ να είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Είναι περίπλοκο και αν κοιτάξετε τις ημερομηνίε θα το διαπιστώσετε. Σκοπός μας είναι να συζητήσουμε και τις ε, εκτελεστικές διατάξεις, την εφαρμογή και εδώ βεβαίως ο χρόνος είναι κάτι που μας απασχολεί. Στην τρίτη διαφάνεια διαπιστώνεται ποια είναι η εφαρμογή αυτής της πρότασης. Πάντα συζητούμε για τα οχήματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εκτός δρόμου, δηλαδή τέσσερις τροχοί. Τα quad και αλλά τα οποία σήμερα ε, είναι αντικείμενα εξαιρέσεων και τα οποία βεβαίως θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο φάσμα της ε, εφαρμογής αυτού του κανονισμού. Θα συζητήσουμε επίσης όλα αυτά τα θέματα στην έκθεσή μας. Κάτι το τελείως διαφορετικό που είναι τα ηλεκτρικά ποδήλατα, μοτοποδήλατα για τα οποία η κατάσταση είναι εξαιρετικά ασαφής. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα πρέπει να γίνει. Υπάρχει σήμερα η ανάγκη για περισσότερη καινοτομία και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε και να προωθήσουμε αυτή την καινοτομία. Ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο είναι βεβαίως η ασφάλεια, το αυτόματο σύστημα φώτων. Αυτό είναι κάτι που το στηρίζουν οι περισσότερες κατηγορίες. Βλέπετε ότι οι οδηγοί μοτοσυκλετών αναφέρονται σε αυτό σαν ένα περιορισμό της ελευθερίας. Επίσης τα συστήματα πέδησης όπως το ABS. Το ABS είναι το σύστημα, προχωρημένο σύστημα πέδησης που ε, μέχρι τώρα υποστηρίζεται από τους περισσότερους καταναλωτές. Θα δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να εξετάσουμε τα διάφορα συστήματα. Σήμερα το απόγευμα θα μιλήσουμε για το σύστημα ABS και τις διάφορες άλλες δυνατότητες τεχνικές που μας προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. Τώρα, όσον αφορά τους ε, προμηθευτές, σήμερα οι μοτοσυκλετιστές ε, θέλουν να χρησιμοποιήσουν ανταλλακτικά τα οποία δεν εμπίπτουν στο φάσμα του κανονισμού αυτού. Και εδώ μας ε, αναφέρουν τον περιορισμό της ελευθερίας. Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κανείς μηχανισμούς που βελτιώνουν τις επιδόσεις των ε, μοτοσυκλετών και των ελαφρών αυτών οχημάτων. Ένα άλλο θέμα, κύριε Πρόεδρε, είναι η εποπτεία και ο έλεγχος της αγοράς. Εδώ πολλά πρέπει να γίνουν. Παρ' όλα αυτά, πολλές προτάσεις ε, έχουν εξεταστεί στα πλαίσια αυτής της έκθεσης και βεβαίως θέλουμε να δούμε τι δυνατότητες έχουμε σήμερα για την καλύτερη εποπτεία και έλεγχο της αγοράς. Ελπίζω με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μπορέσουμε να προτείνουμε διάφορες ε, δυνατότητες για ένα καλύτερο έλεγχο της εσωτερικής αγοράς. Μια πολύ σημαντική πρόκληση είναι το περιβάλλον. Θα πρέπει εδώ να δούμε λοιπόν τους ρήπους, τις εκπομπές και να δούμε ποιες είναι αυτές οι προδιαγραφές που θα επικρατήσουν. Το θέμα της διάρκειας ζωής, της διάρκειας ζωής ενός οχήματος, όσον αφορά βεβαίως στις εκπομπές ρήπων. Κάποιοι προτείνουν επίσης ένα διαφορετικό τρόπο υπολογισμού των εκπομπών ανά ώρα, ανά, ε, σύμφωνα με τη χιλιομετρική απόσταση και βεβαίως το θέμα της εφαρμογής και της αξιοπιστίας των ελέγχων. Αν δηλαδή η προσέγγιση που έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα θα πρέπει να ανανεωθεί βάσει της νέας τεχνολογίας. Αυτά είχα να σας πω. Αυτά είναι τα εισαγωγικά μου σχόλια. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι έχουμε πολλούς οι οποίοι μας ακούν και ίσως όλοι δεν γνωρίζουν όλα τα ακρονίμια. Τι σημαίνει παραδείγματο χάρη OTC ή αλλά αρχικά τα οποία εμείς ευρέως χρησιμοποιούμε και τα γνωρίζουμε. Οι μηχανισμοί παραδείγματο χάρη θα πρέπει ίσως να εξηγούμε λίγο αυτό το λέμε. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Και όπως ξέρετε έχουμε τρία διαφορετικά τμήματα της ακρόασής μας που αφορούν ε, τρει ε, βασικού τομεί τη πρόταση. Θα μιλήσουμε καταρχά για την ασφάλεια, μετά για τι περιβαλλοντικέ επιδόσεις και μετά για θέματα εφαρμογή, που ε, συμπεριλαμβάνουν θέματα χρονοδιαγράμματο, εποπτεία τη αγορά, εφαρμογή κτλ. Έχουμε δύο μιλητέ, δύο εμπειρογνώμονες σε κάθε τμήμα. Κάθε ένα από εσά έχει το πολύ 8 λεφτά. Έχω αυστηρέ οδηγίε από την ΙΜΚΟ. Επομένω, θα χτυπήσω το σφυράκι μου έντονα, αν ξεπεράσετε αυτό το χρόνο. Στο πρώτο τμήμα ε, θα μιλήσουμε για την ασφάλεια. Θα ακούσουμε τον κύριο Λούκα Πασκότο, που είναι Διευθυντής Κινητικότητας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, της ΦΙΑ, που είναι η μεγαλύτερη οργάνωση για τα αυτοκίνητα στον κόσμο και εκπροσωπεί εκατοντάδες χιλιάδες, θα μας πει πόσες εκατοντάδες χιλιάδες μέλη έχει αυτή η ΦΙΑ και μετά ο Πατρίς Ασεντέλ της ε, βασιλικής οργάνωσης ε, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών. Ο κύριος Βιν Βαντενκάμπ είναι μέλος αυτής της ε, οργάνωσης, ενεργό μάλιστα μέλος. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Λούκα Πασκότο για να μας παρουσιάσει τη δική του παρουσίαση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας μιλήσω ε, για τη δική μου εμπειρία, ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο, άρα δεν θα σταθώ στις δύο πρώτες διαφάνειες, εκπροσωπώ τους χρήστες, τους μοτοσυκλετιστές. Ε, χρήστες δηλαδή μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών. Μιλάω λοιπόν εξ ονόματος αυτών των ανθρώπων. Ξεκινάμε με αυτή τη διαφάνεια. Είμαστε πεπισμένοι ότι συχνά ο οδηγό είναι υπεύθυνο για το ατύχημα. Αυτό είναι αλήθεια, εν μέρη. Θα πρέπει να δούμε όμως ε, κατά πόσο μπορούμε να προωθήσουμε ένα σύστημα ασφάλεια, ε, εστιάζοντας και στο χρήστη και στο όχημα και στην ε, υποδομή του δρόμου. Φυσικά, ε, το ατύχημα οφείλεται και στο, σε λάθο ανθρώπινο, αλλά ένα σύστημα ε, μετριάζει αυτό το λάθος, ένα σύστημα κατάλληλο ασφάλεια, μετριάζει αυτό το, το λάθος. Και έχουμε λιγότερα ατυχήματα, κυρίως θανατηφόρα. Να μια σειρά από στοιχεία που μπορούν να συντελέσουν για να αποφύγουν, αποφύγουμε τα μοιραία ατυχήματα. Φυσικά, η εμπειρία και η κατάρτιση και η εκπαίδευση είναι βασικό εργαλείο για οποιοδήποτε οδηγό, αλλά και σωστή σηματοδότηση ε, σε σταυροδρόμια που είναι ψηλού κινδύνου. Βοηθούν τους οδηγούς. Επίσης, ε, η υποδομή, η χερσαία υποδομή, η υποδομή των δρόμων. Επίσης, τεχνικές πληροφορίες είναι τμήμα του συστήματος ασφάλειας, θα το συζητήσουμε αργότερα. Θα πρέπει ε, να υπάρχει πρόσβαση σε τεχνικές πληροφορίες, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τους χρήστες και να έχουμε αποτελεσματικά οχήματα στο δρόμο. Και βεβαίως το τελευταίο στοιχείο, καθώς ε, βελτιώνεται η τεχνολογία. Μην ξεχνάμε ότι τα μοιραία. Έχουμε το ABS βέβαια στο τέλος, Μην ξεχνάμε ότι τα μοιραία ατυχήματα γίνονται όταν κάποια από αυτά τα στοιχεία του συστήματος ε, δεν, δεν λειτουργεί, εν πάση περιπτώσει. Πάμε σε αυτή τη διαφάνεια θα σας εξηγήσω ότι οι οδηγοί δεν είναι ίδιοι παντού στην Ευρώπη. Αριστερά έχουμε τους Ιταλούς, δεξιά έχουμε τους Γερμανούς. Αριστερά έχουμε μια μεσογειακή χώρα και δεξιά μια βόρεια χώρα. Ε, χρησιμοποιούν διαφορετικά οχήματα, άλλους κινητήρες. Αριστερά θέλουν να τα χρησιμοποιούν για περισσότερη κινητικότητα στις πόλεις και δεξιά για λόγους ψυχαγωγίας. Επόμενη διαφάνεια. Βλέπουμε ποιες είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου. Θα δείτε στο έγγραφο διάφορες εξηγήσεις ε, για αυτή την έννοια. Δεν θέλω να σταθώ τώρα εδώ. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια, στην ε, δυνατότητα που μας δίνει η τεχνολογία και κυρίως το ABS, το Anti-Lock Braking System. Ε, η τεχνολογία μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο, ειδικά στα στις μοτοσυκλέτες, υπόσχεται πολλά, με βάση κάποιες δοκιμές ε, ε, οργανώσεων καταναλωτών που έγιναν κυρίως από γερμανικές και ιταλικές οργανώσεις, το ABS ε, εξασφαλίζει και καλύτερη σταθερότητα κατά την πέδηση και μείωση της απόστασης που διανύεται κατά την πέδηση. Και θεωρείται ότι μπορεί να μας οδηγήσουν να αποφύγουμε ή να μετριάσουμε τα μοιραία ατυχήματα. Φυσικά το ABS δεν σημαίνει αυτόματα ασφάλεια. Μόνο αν έχουμε πρακτική και γνωρίζουμε πώς να τα χρησιμοποιούμε το ABS, εξασφαλίζεται η ασφάλεια. Επίσης, να είμαστε ξεκάθαροι. Ο πρόεδρος είπε ότι ABS, μιλάμε για το Anti-Lock Braking System. Ε, καλύπτουμε συστήματα δηλαδή τα οποία μπορούν να εμποδίσουν το μπλοκάρισμα, το κλείδωμα θέλετε της ρόδας ε, κατά την ε, πέδηση. Ε, η συντονισμένη και η σύνθετη και το σύνθετο σύστημα απέδηση είναι καλά συστήματα, αλλά δεν έχουν τα ίδια πλεονεκτήματα με το ABS. Είναι άλλα πράγματα. Τώρα, βλέπετε πόσα συστήματα ABS έχουμε στην Ευρώπη, πού χρησιμοποιούνται. Σε μικρότερους κυβισμούς, κάτω από 250 cc, ε, σπάνια βρίσκουμε ε, ABS, είναι δυνατότητα που την αγοράζουμε έξτρα προχωρούμε. Είναι θέμα κόστους βέβαια. Παραδείγματο χάρη Ιταλή. Στην Ιταλική αγορά, που είναι μια από τις πιο σημαντικές, ε, έχουμε πάρα, πολλά, πάρα πολλές μοτοσυκλέτες, διεισδύει λίγο-λίγο το ABS, αλλά υπάρχει ένα θέμα κόστους. Θα έπρεπε κανονικά να βάζουμε το ABS και ταυτόχρονα υπάρχει μείωση της τιμής. Θα πρέπει επίσης ε, να εκπαιδεύουμε τους οδηγούς ε, στη χρήση του ABS. Υπάρχει ένα πρόβλημα ενημέρωσης ε, πρέπει να ενημερώνονται καλύτερα οι καταναλωτές για τα ωφέλη του ABS. Περιπίν. Βλέπουμε ε, ότι έχουμε μια μείωση κατά μέσο όρο της απόστασης πέδησης κατά 25%. Ε, στο κέντρο δοκιμών στη Γερμανία κάναμε αυτές τις δοκιμές και προέκυψαν αυτά τα αποτελέσματα, όπως βλέπετε. Επίσης με το ABS αποφεύγουμε ή μειώνουμε τις, τα ατυχήματα, τις συγκρούσεις ε, σε διάφορα σταυροδρόμια. Με διάφορες, ε, υπάρχουν διάφορες έρευνες που δείχνουν ότι είναι αποφελές το ABS. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε μία έρευνα για ατυχήματα στην Ιταλία του, το 2008. Θα είχαμε αποφύγει 23% ατυχήματα δηλαδή πάνω από 200 τόσα από τα 1150. Αυτά τα νούμερα επιβεβαιώνονται και από ανάλυση που έχει γίνει στη Γερμανία. Ε, ανάλογο μερίδιο μείωση των ατυχημάτων έχουμε και εκεί. Θα πρέπει να τα διερευνήσουμε περισσότερο αυτά τα αποτελέσματα, ε, δεδομένου της, ε, δεδομένης της μικρής διείσδυσης του ABS στην αγορά. Δεν θα πρέπει όμως να υποτιμούμε τα ωφέλη του ADS, γιατί υπάρχουν και άλλες αναλύσεις που δείχνουν και συγκεκριμένα μια βρετανική ανάλυση ότι τα αποτελέσματα είναι ακόμα πιο θετικά. Πάμε τώρα στις συστάσεις. Επιβεβαιώνουμε ότι η καλή α, κατάρτιση ε, μια εκστρατεία ενημέρωσης. Αυτά είναι στοιχεία εκ των ΟΝΟΚΑΝΕΦ για, την, για τους οδηγούς. Υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες, αλλά το πιο ασφαλές σύστημα είναι το ABS, το Anti-Lock Braking System, το σύστημα απεμπλοκής. Και πιστεύουμε ότι τα μηχανές που είναι πάνω από 125 κυβικά θα πρέπει να, να έχουν οπωσδήποτε, μάλλον το συντομότερο δυνατόν, ABS. Τι, τι σημαίνει αυτό το συντομότερο δυνατόν. Ο ΙΕ ζήτησε από τα κράτη-μέλη να σημειώσουν σημαντική πρόοδο την επόμενη δεκαετία. Το 2017 το ABS σημαίνει α, ότι δεν θα το έχουμε στην αγορά έτσι μαζικά πριν το 2018-2019. Εμείς προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τους οδηγούς, πιστεύουμε ότι θα σημειώσει τη διαφορά σε θέματα ασφάλειας που αφορά αυτή την ε, πολύ εκτεθειμένη ομάδα οδηγών. Σας ευχαριστούμε πολύ για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Υπάρχουν κάποια σημεία που θα πρέπει να αποσαφινιστούν ε, για τους ενδιαφερομένους υστερότερα. Στη συνέχεια, ο κύριος Εσεντέρφτ καλείται να μας δώσει την παρουσίασή του από την Ένωση Μοτοσυκλετιστών της Ολλανδίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ζητήσω να ευχαριστήσω για την δυνατότητα παρουσίασης. Η Ένωση Μοτοσυκλετιστών ε, Ολλανδίας τιμάτε με τη συμμετοχή σε αυτή την ακρόαση. Έχουμε μακρά πείρα. Θα ήθελα να ξεκινήσω δίνοντας μια ιδέα του τι είναι το ABS και τι συνεπάγεται. Και θα αναφερθώ σε κάποια σημεία στη συνέχεια που αφορούν την έκθεση Φαντεκάμψ. Βλέπουμε ε, ότι υπάρχουν τα θέματα και των αναβατών. Το ABS είναι η προτίμησή μας σε μεγάλο βαθμό. Σίγουρα συνιστούμε το ABS δεν θα πηγαίναμε τόσο μακριά ώστε να είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση του ABS, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε τα ωφέλη, όχι μόνο για τις μεγάλες κατηγορίες μοτοσυκλετών, αλλά και για τις ελαφρότερες κατηγορίες. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια θετική λύση, εφόσον θα είχε ευρύτερη χρήση. Και αναφέρθηκε και στην εισαγωγή σε σχέση με ειδικά οχήματα enduro και ε, ειδικά ταχαία οχήματα θα ε, έπρεπε να ζητηθεί να εγκαθίστανται αυτοί, να αυτός ο εξοπλισμός και σε αυτά όμως αναφέρθηκε επίσης ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διευκόλυνση Είμαστε υπέρ του να διατηρηθεί ο εξοπλισμός αυτός εκεί όπου δεν υφίστανται ξεχωριστά ζητήματα. Ξέρουμε από κάποιες εκθέσεις και μελέτες ότι υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις λόγω της τεχνικής κατάστασης ή εξοπλισμού ενός οχήματος Υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά το επίπεδο ε, ηχητικής ε, όχλησης, ε, επίπεδο θορύβων. Για το ABS όμως θα πρέπει να κατανείμουμε σε δύο κατηγορίες τον εξοπλισμό. Δεν ε, ελέγχεται η το απότομο φρενάρισμα και θα πρέπει να μπορεί κανείς με ιδιαίτερα δυνατό τρόπο να μπορέσει να φρενάρει ώστε να είναι ελέγξιμη η πορεία του ε, δικύκλου. Σε όλες τις ε, περιπτώσεις αυτές ε, λέμε πόσο σημαντικό είναι να διδάσκονται, να καταρτίζονται οι αναβάτες πώς να φρενάρουν σωστά ώστε να χρησιμοποιούν ε, τις δυνατότητες του ABS ε, και να ε, μπορούν να υποφεληθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πρέπει να έχουν ειδικά μαθήματα, προηγμένα μαθήματα αξιολόγησης κινδύνου, να προλαμβάνουν την κατάσταση δηλαδή, να προδικάζουν, να κρίνουν προτού χρειαστεί ένα απότομο φρενάρισμα ανάγκης. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε την έκτη αίσθηση στους ε, αναβάτες, ε, να εξετάζουν τους κινδύνους που μπορεί να παρουσιαστούν, να κρίνουν και να δουν πού ελοχεύουν κίνδυνοι σε ε, μία οδό και να προλάβουν μία επικίνδυνη επικίνδυνη κατάσταση. Δυστυχώς έχουμε παραδείγματα καθημερινά και βλέπουμε ότι υπάρχει υψηλό ποσοστό ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται οι μοτοσυκλετιστές σε σχέση με τα χιλιόμετρα που καλύπτουν για παράδειγμα ε, σε σχέση με εμπλοκή και οχημάτων αυτοκινήτων ε, στα ατυχήματα αυτά στα οποία εμπλέκονται και οι μοτοσυκλέτιστες. Είναι και θέματα προτεραιότητας με βάση τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Όμως θα πρέπει έγκαιρα να μπορεί κανείς να μειώνει ταχύτητα, να αφήνεται αρκετή απόσταση με το προπορευόμενο όχημα για να μπορεί κανείς να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει ένα επίγον ε, περιστατικό διδάσκουμε σε ειδικά μαθήματα τους αναβάτες να μπορούν να κρίνουν το τι τεκταίνεται και πώς θα πρέπει να αξιολογούν τους κινδύνους για να αντιδρούν έγκαιρα. Οι αναβάτες έχουν έτσι καλύτερες προοπτικές ε, να οδηγήσουν με ασφάλεια και ε, να μην κινδυνεύσουν. Προσπαθούμε να διδάξουμε τους ε, αναβάτες. Έχουμε και κάμερες που βρίσκονται ε, εγκατεστημένες ε, στο, στη μοτοσυκλέτα τους για να δουν και να αξιολογήσουν ποιοι ήταν οι κίνδυνοι και πώς αντέδρασαν. Προσπαθούμε σε ένα κύκλο ε, μαθημάτων να καταρτήσουμε αυτούς τους οδηγούς όταν προσέρχονται σε εμά κατά τη διάρκεια αυτών των μαθημάτων κατάρτισης μπορούν να εξοικειωθούν με αυτές τις εισαγωγικά δύσκολες ή επικίνδυνες καταστάσεις και να αποκομίσουν ωφέλη. Και έχουμε και επιχορηγήσεις, 200.000 ε, για παράδειγμα ευρώ ήταν για εφέτος και φυσικά είναι επιθυμές να γνωρίζουν οι οδηγοί ποιοι είναι οι κίνδυνοι ώστε να είναι σε θέση να τους αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικό τρόπο. Ο ανθρώπινος παράγοντας, και το είδαμε αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικός, διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Και ο εξοπλισμός του οχήματος είναι ένα άλλο ε, σκέλος. Όμως ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο πιο σημαντικός όταν πρόκειται για την μείωση των κινδύνων και των ατυχημάτων. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την εισαγωγή σας και τώρα θα ξεκινήσει η συζήτηση με παρεμβάσεις από τους ευρωβουλευτές και θα συμμετάσχουν όλοι και ο κύριος Φαντεγκάμ, ο εισηγητής μας. Θέλω να χαιρετήσω και τον κύριο Βεν Λάγκα που είναι μέλος της Επιτροπής Βιομηχανίας και που θα εκπροσωπήσει τον α, εισηγητή των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Είσαστε και εσείς μοτοσυκλέτσις καθ' ό,τι γνωρίζω και ο κύριος Μάντας είναι εδώ επίσης και άλλοι συνάδελφοι και εγώ είμαι σκιώδης εισηγητής ε, για λογαριασμό της ομάδας μου θα προσκαλέσω τους συναδέλφους ευρωβουλευτές να διατυπώσουν ερωτήσεις λοιπόν προς τους ομιλητές. Ίσως ας ξεκινήσουμε λοιπόν, θα επανέλθω στον εισηγητή προς το τέλος αν επιθυμείτε, για να ξεκινήσουμε τώρα. Εσείς κύριε να ξεκινήσετε με τις ερωτήσεις παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο κύριος Λάνε. Νομίζω η αποτελεσματικότητα του ABS είναι αδιαφυσβήτη. Εγώ ο ίδιος ε, είμαι της πρόεδρε. Και εδώ και 9 χρόνια οδηγώ τέτοια, τέτοιες μοτοσυκλέτες με συστήματα ABS ε, anti-blocking system και έχει αυξήσει αυτό την ασφάλεια σημαντικά. Όταν κάνουμε λόγο τώρα για υποχρεωτική εισαγωγή αυτού του συστήματος τίθενται δύο ερωτήματα για μένα. Αφενός, ακριβώς όταν έχουμε μικρότερου κυβισμού μοτοσυκλε... Ε, μοτοσακό ή ε, σκούτερ πρέπει να δούμε τι γίνεται σε σχέση με την προσιτή όσον αφορά την τιμή ε, δυνατότητα εξοπλισμού με το ABS και να δούμε τι γίνεται σε σχέση με την πίεση για τον ανταγωνισμό για αυτά τα μικρότερα οχήματα. Κάποιος μπορεί να μας πει για παράδειγμα τι γίνεται σε σχέση με την εξέλιξη των τιμών, την αύξηση των τιμών με τα μεγαλύτερα οχήματα όταν μέχρι το 2017 θα έχουμε την υποχρεωτική εισαγωγή του ABS, η διείσδυση στην αγορά του ABS θα είναι πολύ καθυστερημένη. Δεν θα ήταν δυνατόν ενδιάμεσα να έχουμε μια ξεκλίμακα σε ε, μια βαθμιδόν ε, εισαγωγή βήμα προς βήμα ε, του ABS στα συμμοτοσυκλέτες ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Φυσικά Έχει σημασία που εφαρμόζεται το ABS. Είναι διαφορετικό για τα μοτοποδήλατα και τα σκούτερ και διαφορετικό για τις μεγαλύτερου κυβισμού μοτοσυκλέτες. Λοιπόν, ο κύριος Μάντες τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν από 25 χρόνια είχα ένα πολύ σοβαρό ατύχημα ενώ οδηγούσα μοτοσικλέτα και άλλαξε τη ζωή μου. Άρα συμφωνώ απόλυτα με αυτά που μας, είπε, μας είπαν οι ομιλητέ από την οργάνωση μοτοσυκλετιστών. Το πρόβλημα συχνά δεν είναι δικό μας των μοτοσυκλετιστών, αλλά των υπόλοιπων οδηγών. Θα πρέπει λοιπόν να γίνονται προσωμιώσει και στους άλλου, καθώς εκπαιδεύουμε και τους άλλους οδηγούς, για να δουν και αυτοί να συνειδητοποιήσουν τι επιπτώσεις έχει η συμπεριφορά τους στους οδηγούς μοτοσυκλετών. Κάτι άλλο. Δεν δείτε; αρκετή προσοχή στα καλάθια, στα παράπλευρα αυτά αυτοκινητάκια των μοτοσυκλετών. Πρέπει να υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές για να βελτιωθεί η ορατότητα στο πλάι. Οι τεχνικές απαιτήσει για τα οχήματα είναι ένα δεδομένο, αλλά χρειαζόμαστε και ένα έξυπνο σύστημα ενημέρωσης, Είδα κάτι σχετικό σε ένα φεστιβάλ για νέες τεχνολογίες που είχα πάει. Πρέπει να είμαστε πρακτικοί για να προβλέψουμε, να προλάβουμε τα ατυχήματα. Κάτι που μου φαίνεται σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν ελάχιστα ευρωπαϊκά όρια ασφάλειας για τα οχήματα και κυρίως τα εισαγόμενα οχήματα, τις εισαγόμενες μοτοσυκλέτες. Γιατί συχνά όταν κατασκευάζονται τα οχήματα εδώ πλήρουν τις προδιαγραφές. Αλλά μοτοσυκλέτες που κατασκευάζονται εκτός ε, Ευρώπης εισάγονται, αλλά δεν έχουν αθέσει τις προδιαγραφές που απαιτούμε εμείς και δημιουργούν προβλήματα στους δρόμους. Για τη συντήρηση τώρα. Θα πρέπει να έχουμε ε, τακτικούς ελέγχους στα, στις μηχανές. Θα πρέπει να έχουμε έτσι μια θεώρηση πιο μακροπρόθεσμη. Θα πρέπει οι μοτοσικλέτες να προσαρμόζονται στην εξέλιξη της τεχνολογίας και να προσαρμόζονται και οι προδιαγραφές λοιπόν, να γίνονται πιο αυστηρές. Για τα ηλεκτρικά οχήματα τώρα, θα πρέπει να δούμε τι λύσεις μπορούμε να βρούμε. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ. Μιλάμε για τον εξοπλισμό ασφάλειας. Έχουμε άλλα δύο πάνελ συζήτησης, επομένως θα επανέλθουμε. Εν πάση περιπτώσει βλέπω ότι δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον. Η κυρία Ρούιλε. Θα ήθελα να αναφερθώ στον πρώτο αγορητή και να ρωτήσω συγκεκριμένα κάτι. Τίθεται το ερώτημα του μεγέθους της μοτοσυκλέτας. Σε ποιο βαθμό αναφέρονται τα θανατηφόρα ατυχήματα με το μεγάλο κυβισμό, την ταχύτητα και ποιο ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίζει το ABS. Είναι ένα θέμα το οποίο ε, σκέφτηκα και πρέπει να απαντηθεί. Το άλλο το οποίο σημείωσα στην έκθεσή σας, είπατε ότι τα περισσότερα ατυχήματα προκαλούνται μέσα σε, στις ίδιες τις πόλεις. Και εδώ υπάρχουν μελέτες σε σχέση με την ε, επίπτωση της επιπτώσης του ABS σε σχέση με την χρήση ε, του, της μοτοσυκλέτας αξίζει και για μικρότερες μοτοσυκλέτες, για μοτοποδήλατα, για παράδειγμα μοτοσακό, να χρησιμοποιείτε το ABS στις πόλεις και σε ποιες περιπτώσεις αυτό θα είχε ωφέλη. Και σε σχέση και για το πώς θα μπορούσε αυτό να έχει επιπτώσεις στο κόστος, πώς θα μπορούσε το κόστος να μειωθεί. Αυτό σε σχέση με τα μικρότερα, με, τις, με, τα μικρότερα οχήματα είναι δεδομένο ερώτημα. Διότι για τα μεγάλα, τις μεγάλες μοτοσυκλέτες το κόστος δεν μπορεί να είναι ο αποφασιστικός παράγοντας. Ευχαριστώ. Έχετε τον λόγο εσείς παρακαλώ. Ο κύριος Ρέπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εδώ δεν είναι μόνο το θέμα της αποτελεσματικότητας και της σημασίας του ABS που δεν θέλω με κανένα τρόπο να αμφισβητηθεί, διότι αναφέρθηκε ούτως ή άλλως ότι είναι μια σημαντική πτυχή υπέρ της ασφάλειας του ABS. Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτά τα οποία συμβαίνουν στα δίκυκλα, αλλά και αυτά τα οποία συμβαίνουν με τους αναβάτες. Και αυτός ο παράγοντας, ο ανθρώπινος παράγοντας διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και θα ήθελα ακριβώς σε σχέση με τους νεότερους μοτοσυκλετιστές να το αναφέρω αυτό. Πιστεύω εκεί υπάρχουν ε, κάποιες νέες ε, καινοτομίες που είναι αναγκαίες ε, για να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Διότι για πολλούς τι συμβαίνει. Είναι εξαιρετικό να έχουν ένα πρώτο, μια πρώτη μοτοσικλέτα που αγοράζουν για να κάνουν το κέφι τους. Πολλοί νέοι. Όμως το ερώτημα είναι μέχρι πού μπορεί να φτάσει κανείς και πώς μπορούν όλα αυτά τα θέματα να ρυθμιστούν νομοθετικά για να προστατεύονται αυτοί οι αναβάτες. Δεν ξέρω τι γίνεται με τις υποπροδιαγραφές ε, επιβολή εξοπλισμών για την ασφάλεια. Όταν αγοράζει κάποιος μια μοτοσυκλέτα εκείνο το οποίο μετρά είναι πώς μπορεί να ελέγξει και να οδηγήσει με ασφάλεια αυτό το όχημα. Σε αυτό τον τομέα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε με προτεραιότητα. Πρόεδρος, θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ υπό τον ρόλο μου ως κοιόδης εισηγητή σε κάποια θέματα με κάποιες ερωτήσεις που θα είχα. Απλά θα ήθελα να επικεντρωθώ περισσότερο στα θέματα της ασφάλειας που βρίσκονται στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια σχετικά καθαρή εικόνα από πλευρά σας ότι είσαστε υπέρ της ένταξης και της χρήσης του ABS για πολλούς λόγους και υποστηρίζονται αυτά, αυτό, αυτά τα αιτήματα από τα τεκμήρια και τις αποδείξεις. Τώρα, σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε σχέση με ένα ε, συγκεκριμένο μέγεθος ε, δικύκλων για την εγκατάσταση του ABS από ένα μέγεθος και πάνω, από ένα κυβισμό και παραπάνω. Τι γίνεται με τα μικρότερα όμως αυτό είναι ένα θέμα. Μια εναλλακτική μορφή συνδυασμού συστημάτων πέδησης ε, θα έπρεπε ίσως να αναζητηθεί που θα οδηγεί στο να αποφεύγεται το μπλοκάρισμα των τροχών. Αλλά επίσης και σε σχέση με την ε, γνώση που έχουν ε, οι μηχανολόγοι και οι υπεύθυνοι για αυτά είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε αυτά τα στοιχεία. Ίσως θα μπορούσε η Επιτροπή να σχολιάσει τα θέματα αυτά γνωρίζοντας σε σχέση με την δυναμική και το βάρος που επιμερίζονται ε, τα δίκυκλα, έχουν τελείως διαφορετική ε, ιδιότητα τα σκούτερ και τα μοτοποδήλατα από ότι οι μεγάλες μοτοσικλέτες έχουν ε, μεγαλύτερη, μεγαλύτερο βάρος σε σχέση με το βάρος του πίσω επιβάτη, στον πίσω άξονα. Και έτσι εδώ υπάρχουν ιδιομορφίες όταν έχουμε την περίπτωση ενός ε, ε, απότομου φρεναρίσματος. Πώς θα μπορούσε να αποφευθεί η αποσταθεροποίηση ενός τέτοιου δικύκλου. Δεν είναι μόνο το θέμα της απόστασης ε, πέδησης, αλλά είναι επίσης και της, η αντιμετώπιση της, του μπλοκαρίσματος σε πρόορη απότομη πέδηση. Υπάρχει ένας ε, τομέας όπου τα μικρά, ε, οι μικρού κυβισμού ε, μοτοσυκλέτες θα μπορούσαν ίσως να επωφεληθούν. Και θα έπρεπε να δούμε αν το 125 κυβικά εκατοστά είναι ένα όριο, μια διαχωριστική γραμμή για το διαχωρισμό δικύκλων που θα μπορούσαν να εξοπλίζονται με το ABS ή όχι. Και σε σχέση με ειδικέ ε, τώρα ε, μοτοσυκλέτες ε, που δεν θα είχαν ABS αλλά που θα έπρεπε όμως να έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικά οχήματα κατά την πέδηση. Θα πρέπει αυτό να το δούμε Επίσης υπάρχουν πολλά χρήσιμα στοιχεία στην έκθεσή σας που δεν είχαμε ε, τον χρόνο να εμβαθύνουμε σε αυτά που αντανακλούν όμως τις ε, διαφορές μεταξύ αστικών περιοχών και άλλων περιοχών. Και υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό θέμα, ε, το θέμα της κατάρτισης. Ωστόσο αυτό θα έπρεπε να αφορά και τους συναδέλφους στην Επιτροπή Μεταφορών που ήταν, είναι περισσότερο δική τους αρμοδιότητα. Αυτή είναι η δική μου παρέμβαση κύριε Φαντερκάμπ, θα θέλατε να αναφερθείτε στα, στις παρεμβάσεις και να σχολιάσετε παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε τον Άγγλο. Πρώτα απ' όλα ως εισηγητής ε, ο εισηγητή αυτό που πρέπει να κάνει είναι να ακούσει πάρα πολύ προσεκτικά, να αφουγκραστεί τι απόψει των πολιτών. Δεν πιστεύω όπως πολλοί ε, άλλοι ότι γνωρίζω τα πάντα. Δεν πρέπει κανείς να νομίζει ότι γνωρίζει τα πάντα. Πρέπει όμως ε, με κοινό νου να λαμβάνονται υπόψη οι απόψει ε, των μοτοσυκλετιστών ε, σε σχέση με τα θέματα ε, της συμπερίληψης του ABS στις μοτοσυκλέτες. Υπάρχει εδώ λοιπόν η πλειοψηφία σε σχέση με τα όσα αναφέρθηκαν που λένε, λέει αυτή η πλειοψηφία ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε το σύστημα ABS στις μοτοσυκλέτες γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Δεύτερο σχόλιο για το χρονοδιάγραμμα. Δεν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία προτού αν δεν προχωρήσει το Συμβούλιο και η Επιτροπή αν δεν προχωρήσουν πιο γρήγορα, δεν επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Λυπούμε που τα πράγματα δεν έχουν επιταχυνθεί, όμως ε, στις συνεδριάσεις πρέπει να επιταχυνθούν περισσότερο οι διαδικασίες. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2017 να ολοκληρώσουμε. Δεν απομένει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Μετά σε σχέση με την ε, ελευθερία ή το περιθώριο που απομένει και το περιθώριο να μπορεί κανείς ε, να ε, λάβει αποφάσεις. Δεν είναι δυνατόν να εξετάζουμε εδώ την πτυχή του του να γίνονται ταχύτερε οι μοτοσυκλέτε με το να πειράζουμε τη μηχανή. Όμως από την άλλη πλευρά υπάρχει προσπάθεια για τα trial και τα enduro να ενταχθούν στον κανονισμό αυτά τα δίκυκλα. Καλό είναι, μπορεί να γίνει αυτό. Από την άλλη όμως πλευρά πρέπει να πούμε να είμαστε προσεκτικοί. Προσέξτε, διότι διαφορετικά α, δεν θα μπορούσαν να ενταχθούν το ABS, να ενταχθούν στο πλαίσιο του ABS. Πρέπει να δούμε ε, ξεχωριστά τα θέματα των εντούρο, για παράδειγμα. Ε, και σε σχέση με τις ερωτήσεις, ε, η παρουσίαση στην σελίδα 4 καθορίζεται η αναλογία μεταξύ κατάρτισης και πείρας με την χρήση ABS για τους αναβάτες. Και διαρωτώ με, αληθεύει δεν είναι σωστό ότι 70% των ατυχημάτων προκαλούνται από τη συμπεριφορά του ίδιου του αναβάτη γνωρίζουμε ότι τα στοιχεία του ADAC, του Γερμανικού Ομίλου Αυτοκινητιστών, οδηγούν στο να μπορεί να πει κανείς ότι μειώνονται τα ατυχήματα αυτά με τη χρήση του ABS. 70 όμως 100 όπως είπαμε των ατυχημάτων προκαλούνται από την ίδια τη συμπεριφορά του αναβάτη. Πολλές φορές αυτό οφείλεται και σε συμπεριφορά των ίδιων των οδηγών αυτοκινήτων από την άλλη πλευρά. Αυτό επαληθεύεται κύριος Εσεντεύτε και μετά στη συνέχεια ο άλλος αγορητής να απαντήσουν και να τοποθετηθούν. Έχετε παρακαλώ τον λόγο. Πιέζει όμως ο χρόνος, έχετε όμως ε, λίγα λεπτά να απαντήσετε κι εσείς παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος ε, στην ε, απάντηση που θα δώσω, διότι οι ερωτήσεις αφορούσαν περισσότερο τον κύριο αριστερά μου παρά εμένα τον ίδιο. Θα ήθελα να αποσαφηνίσω ένα συγκεκριμένο θέμα. Ο κύριος εισηγητής Φαντεν Κάμπς είπε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν ίσως εξαιρέσεις για τα, τις μοτοσυκλέτες εντούρο. Εντάξει, όμως να λάβουμε υπόψη και τις μετακινήσεις διότι είναι σημαντικό να περιγράφεται η αναλογία που υπάρχει σε σχέση με τα ίδια τα αυτοκίνητα πολλά ατυχήματα οφείλονται ακριβώς στην αντίδραση στη συμπεριφορά των οδηγών αυτοκινήτων και θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί αν είχε ο άνθρωπος στο τιμόνι, στο αυτοκίνητο, ο οδηγός του γιώταχη αντιδράσει διαφορετικά. Εδώ όμως βλέπουμε το θέμα της ε, απρόβλεπτης αντίδρασης ε, των ε, οδηγών στις κάτω χώρες στην Ολλανδία, αλλά αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και αλλού. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι γενικά οδηγούν 3 ή 4 χιλιόμετρα το χρόνο, από τον Απρίλιο ως τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο κλείνονται οι μοτοσυκλέτες στα γκαράζ. Και έτσι δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για την ε, συλλογή μεγάλη συσσόρευση μεγάλης ε, πύρας. Χρειάζονται λοιπόν μαθήματα, κατάρτιση, διαρκής θα έλεγα επιμόρφωση για να μπορέσουν να συσσωρεύσουν πύρα, να αυξηθεί η ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα της ασφάλειας. Και φυσικά το ίδιο ισχύει και για τα οχήματα, τα ΙΟΤΑΧΗ, που και η δική του συμπεριφορά αφορά και έχει επιπτώσεις στα δίκυκλα και στους οδηγούς δικύκλων. Σας ευχαριστώ. Πασκότο. Σύνθετες οι ερωτήσεις, θα προσπαθήσω να κάνω κάποια σχόλια και μετά στη διάθεσή σας. Ε, χρειαζόμαστε πιο ποιοτικά στοιχεία και για την ασφάλεια και για τα τροχαία ατυχήματα. Θα πρέπει να, να καταλάβουμε τι συμβαίνει στο δρόμο, θα πρέπει να κάνουμε εκτιμήσεις για τα ωφέλη που μπορεί να μας δώσει η τεχνολογία με βάση την έρευνα που έχει γίνει μέχρι στιγμής. Για το κόστος, νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε μια ανάλυση κόστους-οφέλους. Δηλαδή κόστο ό,τι αφορά την υγεία, ό,τι αφορά τη συντήρηση των οχημάτων, τη συντήρηση της υποδομής και πρέπει να τα δούμε όλα αυτά πριν εισαγάγουμε μια σημαντική τεχνολογική αλλαγή. Παραδείγματο χάρη, υπάρχουν διάφορα εξαρτήματα ας πούμε, που στην αρχή ο κατασκευαστής δεν θέλει να εντάξει, αλλά τελικά είναι κλασικά πια ε, και λόγω ανταγωνισμού στην αγορά. Τώρα για αυτό το ποσοστό των 70% ατυχημάτων λόγω της συμπεριφορά των οδηγών. Θα πρέπει οι οδηγοί να είναι σε θέση να λάβουν τη σωστή απόφαση. Εγώ θα ήθελα να σκεφτούμε μέσα στα πλαίσια ενός ασφαλούς συστήματος. Γιατί αν δεν έχουμε καλή κατάρτιση ας πούμε, α, ναι, λάθος του οδηγού είναι, αλλά τελικά το όλο σύστημα χωλαίνει. Ε, νομίζω ότι όλο το σύστημα χάνει, ας πούμε, αν οι οδηγοί α, δεν συμπεριφέρονται με σωστό τρόπο. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ας πάμε λοιπόν στην επόμενη ενότητα. Βεβαίως αν θέλετε να σχολιάσετε ή να πάρετε το λόγο μπορείτε να μου το πείτε. Περνάμε τώρα στο περιβάλλον, στις περιβαλλοντολογικές πτυχές. Έχω δύο ειδικού που θα μας μιλήσουν για το θέμα αυτό. Είναι μεγάλη ευχαρίστηση που μπορούμε να καλωσορίσουμε τον Μπερτχό Ολιβίε Dicreux από την Γαλλική Υπηρεσία Περιβάλλοντος Ενέργειας και θα μας μιλήσει για τις περιβαλλοντολογικές επιδόσεις των οχημάτων, πώς μπορεί να υπάρξει έλεγχος των εκπομπών με καταλήτες. Ο κύριος Ντικρύ θα μας μιλήσει πρώτος και κατόπιν ο κύριος Μπρέσοτ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσουμε καταρχήν για τα δίκυκλα, τα μοτοποδήλατα, τις μοτοσυκλέτες, αλλά και τις επιπτώσεις των ελαφρών οχημάτων επί του περιβάλλοντος, δίνοντας κάποια παραδείγματα. Τα συμπεράσματα στο οποία έχουμε φτάσει φαίνονται από τα στοιχεία που δίνουμε. Αυτά όλα είναι τα αποτελέσματα. Στην αριστερή πλευρά βλέπετε την κατανάλωση Καψίμων και δεξιά τις εκπομπές με την παρουσίαση των διαφόρων κατηγοριών, δικύκλων και ελαφρών οχημάτων που έχουμε πάρει σαν αναφορικές κατηγορίες. Βλέπετε εδώ ότι μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα μηχανοκίνητα δίκυκλα καθώς και η κατανάλωσή τους. Έχουμε τις συγκεκριμένες τιμές χωρίς υψηλή τεχνολογία, τις κατηγορίες low cost και τις επιπτώσεις επί του περιβάλλοντος. Μεγαλύτερα μηχανοκίνητα δίκυκλα για την καθημερινή χρήση. Βλέπετε τα αποτελέσματα, δεν είναι κάτι που μας ξαφνιάζει. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε το WMTC, τον κύκλο δοκιμών και την κατανάλωση. Μπορείτε να διαπιστώσετε ότι η κατανάλωση καυσίμων εδώ είναι πολύ κοντά στην χρήση την οποία έχουμε συγκρίνει και βεβαίως με τις μετρήσεις και τις δοκιμές που έγιναν στα Euro 3. Ακριβώς το ίδιο βλέπετε σε αυτή τη γραφική παράσταση, αφορά όμως η μέτρηση εδώ της εκπομπές διοξιδίου. Στην πραγματική χρήση των οχημάτων αυτών και το WMTC είναι πολύ πιο κοντά στις πραγματικές τιμές σε σχέση με τη διαδικασία Euro 3 σε μια χρήση εντός των αστικών περιοχών και εκτός των αστικών περιοχών. Μετρήσαμε 11 διαφορετικές περιπτώσεις δικύκλων με τις μετρήσεις Euro 3 και βλέπετε εδώ τις οριακές με την κόκκινη διακεκομένη γραμμή. Τι παρατηρήσεις μπορούμε να κάνουμε εδώ. Ότι μεταξύ του WMTC και του Euro 3 υπάρχει κοινή παρουσίαση αποτελεσμάτων αλλά σε πολύ χαμηλές αποστάσεις χιλιομετρικές πέφτουν οι τιμές, είμαστε κάτω από τα ανώτερα όρια. Τρεις κατηγορίες ξεπερνούν και όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου και τις άλλες εκπομπές, αυτές τις ανώτατες τιμές, και αυτό βεβαίως πρέπει να οφείλεται κυρίως σε τεχνικούς λόγους, είτε διότι βρίσκονται στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, Εκτός από αυτές τις κατηγορίες, πρόκειται για κατηγορίες οχημάτων που λειτουργούν με ψεκασμό καυσίμων. 225 κυβικά και κυρίως οι άλλες κατηγορίες είναι 125 κυβικά. Χαμηλές εκπομπές στην αριστερή δηλαδή και κάτω γωνία της γραφικής παράστασης είναι κυρίως ε, ελαφρά οχήματα, δίκυκλα, μοτοποδήλατα, χαμηλού κυβισμού είτε πολύ υψηλής τεχνολογίας, δηλαδή πιο ακριβά οχήματα. Όσον αφορά το OBC, βλέπουμε ότι κάποιες κατηγορίες ξεπερνούν τις ανώτατες τιμές. Τα αποτελέσματα αυτής εδώ της μέτρησης είναι όσον αφορά τις διάφορες κατηγορίες εκπομπών και ρήπων, τρεις κατηγορίες ρήπων. Στην κόκκινη γραμμή βλέπετε ότι υπάρχουν οι αντιστοίχες τιμές με το Euro 3 με, τις, ε, τα πρότυπα Euro 3. Αριστερά είναι τα οχήματα 125 κυβικών και στην δεξιά πλευρά τα οχήματα diesel για τις εκπομπές ε, οξυδίων του αζότου. Θα πρέπει σε γενικές γραμμές να παρατηρήσουμε ότι τα δίκυκλα μηχανοκίνητα βάσει των μετρήσεων ε, Euro 3 έχουν εξαπλάσιες εκπομπές σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες οχημάτων. Θα ήθελα επίσης για να μην καθυστερήσω να, ξεπεράσω, να περάσω στην ε, μεθεπόμενη διαφάνεια Βλέπετε εδώ την σύγκριση για τις εκπομπές οχημάτων 125 κυβικών με κόκκινο και με μπλε το WMTC Euro 1 και 2 την πρόταση δηλαδή που εξετάζουμε εδώ και θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι μοτοσυκλέτες 125 κυβικών εκπέμπουν τόσο πολλούς ρήπους και γιατί θα ήταν πολύ πιο Θα πρέπει με αυτόν τον τρόπο και με τους καταλήτες να μειωθεί η εκπομπή ρήπων σε αυτά τα μηχανήματα. Θα ήθελα επίσης να πω ότι στη Γαλλία οι μετρήσεις μας έδειξαν ότι η πραγματική χρήση και η χρησιμοποίηση αυτών των ε, νέων τεχνολογιών θα μειώσουν σημαντικά και την ηχορύπανση αλλά και τις εκπομπές και υπάρχουν αυτοί οι εξοπλισμοί ήδη στην αγορά Είδαμε επίσης ότι και για την κατανάλωση καυσίμων τα αποτελέσματα είναι καλύτερα. για τα καινούρια μηχανήματα. Και βλέπουμε βεβαίω ότι τα αποτελέσματα είναι πολύ διαφορετικά και αυξάνονται στην πραγματική χρήση. Είμαστε λοιπόν υπέρ των προτάσεων. Θεωρούμε ότι με την WMTC τα αποτελέσματα βελτιώνονται και όσον αφορά τις εκπομπές ε, διοξιδίων του άνθρακα, αλλά και όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμων και θα πρέπει να προσφέρουμε τη δυνατότητα χρησιμοποίησης αυτών των τεχνολογικών δυνατοτήτων. Ξέρουμε σήμερα την μεγάλη σημασία των μηχανοκίνητων δικύκλων σε αστικά κέντρα και θα πρέπει να μπορέσουμε να συγκρίνουμε πραγματικά τα αποτελέσματα αυτής της κατηγορίας οχημάτων με αυτής των αυτοκινήτων. Σας ευχαριστώ πολύ, λέω. Να ξεκαθαρίσουμε τα εξής ότι το WMTC είναι ο κύκλος δοκιμών ε, που γίνεται στον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Είναι μία σειρά από δοκιμές που υφίσταται η μοτοσικλέτα για να δούμε πώς χρησιμοποιείται, με ποιο τρόπο χρησιμοποιείται συνήθως, όταν είναι κρύα και τα λοιπά, σε διάφορες φάσεις. Αυτό το λέω για τους αδαείς που δεν γνωρίζουν ε, τα της μοτοσυκλέτας. Κάτι άλλο που ξεκαθαρίστηκε νομίζω καθοδόν, αλλά είναι σημαντικό για τις μετέπειτα συζητήσει μας, είναι ότι αν κατάλαβα αυτά που είπατε, ειδικά για τις μικρές μηχανός, μηχανές υπάρχουν πολλές διαφορές στις επιδόσεις. Ε, λόγω της φύσης των δοκιμών, λόγω του τρόπου που λαμβάνουν χώρα αυτές οι δοκιμές. Ε, Μπορεί δηλαδή ας πούμε, ε, να έχουμε τελείω διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με το αν έχουμε πειράξει ας πούμε, μία μηχανή ή όχι. Ε, σωστό είναι αυτό. Ναι. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που είπατε για τον κύκλο δοκιμών. Πρέπει να είναι ο κύκλος δοκιμών να γίνεται ε, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική χρήση της μοτοσυκλέτας, τη χρήση στην πραγματική ζωή. Παραδείγματο χάρη, οι ιδιοκτήτε μοτοποδηλάτων, α πούμε, ε, παίζουν πολύ με, τους... με τα καρμπιρατέρ. Παραδείγματο χάρη με τα πενιντάρια, με τα 50 κυβικά. Παίζουν πάρα πολύ. Οπότε αυτό είναι θέμα. Ε, τι γίνεται τώρα με τους καταλήτες, ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Καλησπέρα κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι που είμαι εδώ, σε αυτή την δημόσια ακρόαση. Θα ήθελα να σα δείξω κάποια αποτελέσματα για τρεις, τρία προγράμματα μετρήσεων που έκανε η AECC, που όπω είπατε στην εισαγωγή σα εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Καταλητών. Βλέπετε τι εταιρείε που είναι μέλη τη AECC, βλέπετε τους λογότυπούς τους, αυτή είναι η βασική εταίροι παίκτε στην Ευρώπη, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των εκπομπών, αναπτύσσουν τεχνολογίε για όλα τα κινητά οχήματα. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Αυτό που κάναμε στο πρόγραμμα δοκιμών των μοτοσυκλετών ε, στην AECC, ε, δοκιμάσαμε πέντε μοτοσυκλέτες, ε, οι τρεις είναι 3 γιούρο. τρία είναι κλασικές ε, ε, μηχανές ε, Ευρώπης ή Ασίας ε, και μία με ειδικέ προδιαγραφές. Ζητώ συγγνώμη που δεν μοιράσαμε τις διαφάνειες. Κάποιο λάθος έγινε, αλλά θα σας μοιράσουμε μετά το κείμενο στο Κοινοβούλιο. Βλέπετε στους πίνακες εδώ τις τεχνικές προδιαγραφές αυτών των πέντε μοτοσυκλετών. τις επιλέξαμε για να είναι αντιπροσωπευτικές του στόλου των μοτοσυκλετών. Όταν δοκιμάσαμε αυτές τις μοτοσυκλέτες, παρατηρήσαμε ότι μερικά από τα οχήματα που δοκιμάσαμε δεν ε, ε, περνάνε τις δοκιμές. Η πρώτη ε, που νοικιάζεται, είναι μηχάνημα που νοικιάζεται, είχαμε κάποιους αισθητήρε οξυγόνου που είχαν πρόβλημα και είχε πρόβλημα η μηχανή. Μετά το διορθώσαμε και νομίζω ότι ε, είμαστε εντός των ορίων εκπομπών. Ε, επίσης είχαμε μία εισαγόμενη μηχανή, ε, μηχανή D. Μάλιστα ε, φέραμε μια εισαγομενη μηχανη μηχανη d μαλιστα φεραμε μια δευτερη γιατι την πρώτη δεν μπορέσαμε να την ευθυγραμμίσουμε τα πρότυπα Euro 3. Στο δεύτερη περίπτωση περάσαμε τα όρια Euro 3 μετά από προσαρμογή που το ζήτησε ο εισαγωγέας. Μετά από αυτές τις ενδιαφέρουσες εμπειρίες λοιπόν, βλέπετε τα γερμανικά δεδομένα για την έγκριση τύπου μέχρι το 2009 ε, για το οξύδιο του ε, αζότου και του σιρογονάνθρακες για το Euro 2, 3, 5 και 6. Αν πατήσετε το κουμπί βλέπετε τις τέσσερις μηχανές, όχι τη, μία μηχανή, βλέπετε τις ε, τέσσερις ευρωπαϊκές μηχανές ε, που είναι ευρωτρία, τις οποίες δοκιμάσαμε. Πάνω είναι οι ειδικέ ε, προδιαγραφές. Δεν είναι σχεδιασμένη αυτή, αυτό το μηχάνημα για να σεβαστεί αυστηρά πρότυπα εκπομπών, αλλά για τις προδιαγραφές των, των καυσίμων είναι ok. Εν συνεχεία, οι τέσσερις μοτοσικλέτες ε, σέβονται τις προδιαγραφές Euro 4. Βλέπετε και την μοτοσικλέτα B που είναι ε, στο επίπεδο των προτύπων Euro 6. Με βάση αυτή τη γραφική παράσταση ε, έχουμε καλή τεχνολογία στην αγορά. Τι άλλο κάναμε στο πρόγραμμα δοκιμών μας. Εξετάσαμε τη διάρκεια ζωής τον εισαγόμενο από την Ασία, της από την Ασία ε, μοτοσυκλέτας Β, είχαμε την αίσθηση ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά. Αυτό το συνέστημα επιβεβαιώθηκε. Γιατί καθώς γερνούσε ε, το όχημα, είδαμε ότι οι εκπομπές μονοξυδίου του άνθρακα μετά από 2.000 χιλιόμετρα ξεπέρασαν το όριο. Και για το οξύδιο, το του αζότου ε, μετά από 5.000 ε, δεν υπάρχουν δηλαδή προδιαγραφές ε, διάρκεια ζωής. Αυτό τι σημαίνει ότι έχουμε μοτοσυκλέτες στην αγορά οι οποίες δεν διαρκούν. Πληρούν τις προδιαγραφές για ένα μικρό χρονικό διάστημα αλλά όχι συνέχεια. Τώρα κάποιες δοκιμές για πρόσφατες ευρωπαϊκές, ευρωπαϊκά μοτοποδήλατα. πέντε ευρωπαϊκά μοτοποδήλατα γύρω δύο. Βλέπετε τις προδιαγραφές αυτών των μοτοποδηλάτων. Ε, είχαμε τέσσερα τετρακίνητα, ένα τετρακίνητο με καρμπυρατέρ, ένα δικίνητο μοτοποδήλατο. Όλες οι, όλα τα μοτοποδήλατα, εκτός από τα ε, τετράτροχα, ε, πληρούσαν τις προδιαθέσεις Euro 2. Η δεύτερη, όμως το δεύτερο μηχανάκι δεν ε, πέρασε το τεστ. Οι άλλες, ε, τα άλλα μηχανάκια λειτουργήσαν καλά. Στο, στη δοκιμή Euro 3 υπολογίζουμε το 30% της εκκίνησης με κρύα τη μηχανή σε σχέση με ζεστή τη μηχανή. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά κρύα ή ζεστή μηχανή. όλα τα αποτελέσματα εδώ δεν δείχνουν δεν υπάρχει διάρκεια. Εδώ έχουμε ε, δεδομένα για την έγκριση τύπου από το 2009. Εδώ βλέπετε ε, αυτό το σύννεφο, τα βασικά δεδομένα δηλαδή, ε, εντάσσονται στο κουτάκι Euro 2. Για το Euro 3 δεν υπάρχει αλλαγή στην στα όρια εκπομπών, απλώ ε, κάνουμε την εκκίνηση με κρύο κινητήρα ή με ζεστό κινητήρα. Ε, επίσης, ε, μερικά δεδομένα είναι στο κουτάκι γύρω 4 και το γύρω 5 είναι πολύ πιο δύσκολο να επιτευχθεί. Εδώ βλέπουμε τα μοτοποδήλατα που δοκιμάσαμε. Υπάρχουν κάποιε δοκιμές εδώ πέρα, ανάλογα οι υδρογονάθρακες, οξύδια του αζότου κτλ. Τέσσερα από τα πέντε μοτοποδήλατα, το τετρα Πετράχρονο είναι οριακό. Τα άλλα όμως πληρούν, θα πληρούν μάλλον τις, τα όρια εκπομπών στο εγγύς μέλλον. Τώρα, υπάρχει μια δήλωση στην πρόταση της Κομισιόν ότι η τελική φάση για την νομοθεσία των, ε, των μοτοσυκλετών είναι η ίδια για το Euro 5 για τα επιβατικά αυτοκίνητα. Κοιτάξαμε λοιπόν τον αριθμό του, τη μάζα του, τον όγκο του δηλαδή, ε, και είδαμε τον κύκλο Euro 3 και τον WMTC. Στην ε, κάτω γραφική παράσταση τα συνοψίζουμε. Βλέπετε τη την σύγκριση ανάλογα μέσα στα, στις και στα επιβατικά αυτοκίνητα. Βλέπετε την το μπλε ιστόγραμμα. Ε, είναι ε, diesel κινητήρας. Ο ένας με φίλτρο και ο άλλος χωρίς φίλτρο. Είναι δύο οι στήλες οι μπλε. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Βλέπετε τα αποτελέσματα για τα μοτοποδήλατα το τετράχρονο μοτοποδήλατο με ηλεκτρονική έγχυση. Ε, βλέπετε τα αποτελέσματα που δίνει. Όλα τα άλλα ε, ξεπερνούν τα πρότυπα των αυτοκινήτων. Αν δείτε τη τα... σωματίδια που εκπέμπουν, έχουμε 3,8 ε, επί 10 στη 12η. Πολύ παραπάνω δηλαδή από τις οριακές τιμές. Τώρα κάποια συμπεράσματα σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν. Υποστηρίζουμε την πρόταση της Κομισιόν, ιδίως στις τελικές φάσεις ε, της πρότασης αυτής. Θεωρούμε ότι οι ενδιάμεσες φάσεις ε, θα μπορούσαν να ενισχυθούν. Οι περισσότερες μοτοσυκλέτες και τα μοτοποδήλατα ε, είναι, σέβονται τα, τις επόμενες φάσεις για τα όρια δοκιμών. κάποια τρίτροχα τώρα έχουν ε, χαλάρα όρια εκπομπών, όπως προτείνει το γύρο 3 και γύρο 4, αλλά δεν υπάρχει τεχνικός λόγος για κάτι τέτοιο, αλλά θα πρέπει να αλλάξει. Για τα μοτοποδήλατα ε, θα πρέπει να υπάρχει καλύτερος έλεγχος του κινητήρα ε, για να κάνουμε, να τις προσαρμόσουμε μετά. Για την, τη σωματιδιακή εκπομπή, αντίστοιχα θέματα. Για τα υβριδικά θα πρέπει να δούμε τις οριακές τιμές με, α, με βάση την τεχνολογία του κινητήρα εσωτερικής κάψης. Εμείς ε, θέλουμε να υπάρχουν οι προδιαγραφές για το διαγνωστικό έλεγχο στον πίνακα ελέγχου και κάποιες προδιαγραφές για τη διάρκεια ζωής. Αυτά ευχαριστώ. Ήμουν πολύ γενναιόδωρος όσον αφορά τον χρόνο μαζί σας για τα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε. Οι περισσότερες ε, παρουσιάσεις ήταν ε, πραγματικά εξαιρετικές. Όμως για να είμαστε σύντομοι είναι σημαντικό γιατί τα όσα αναφέρθηκαν με τα θέματα για την ε, ε ανθεκτικότητα είναι και αυτά σημαντικά. Αν συνάδελφοι έχουν ερωτήσεις ε, που θα ήθελαν να διατυπώσουν τώρα, αλλιώς να περάσουμε στην επόμενη φάση. Κύριε Λάγκα, θέλετε να ρωτήσετε κάτι πολύ σύντομα παρακαλώ, πολύ σύντομα. Παρακαλώ. Ναι, ίσως απλά και μόνο το θέμα του συνδυασμού της ε, από κοινού συνδυαστικής προσπάθειας των κλιμάκων 5 και 6. Προφανώς η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ ώστε κάποιες μοτοσικλέτες να προσεγγίζουν το επίπεδο 6, Euro 6. Έχει νόημα να έχουμε μια ενδιάμεση κλίμακα όσον αφορά την βιομηχανία καταλυτών για μια ενδιάμεση κλίμακα. Μια και κάτι τέτοιο, μια ολόκληρη σειρά κόστους ε, και δαπανών ε, για την βιομηχανία θα προκαλούσε. Δεν είναι σκόπιμο να πούμε συγχωνεύονται οι κλίμακες 5 και 6 σε μια ενιαία βαθμίδα και όσον αφορά τα μοτοποδήλατα, τα μοτοσακό, η μόνη καλή επίδοση ήταν με τον τετράχνο κινητήρα μοτοποδηλάτου. Βλέπετε στο μέλλον κάποιες προοπτικές για τους δίχρονους κινητήρες, ε, για τους ε, κινητήρες μοτοποδηλάτων που είναι ε, δίχρονοι. Ευχαριστώ πολλές ερωτήσεις. Κάποιος που θα ήθελε να απαντήσει ή να τοποθετηθεί, εσείς θα θέλατε να αναλάβετε την απάντηση, ίσως κύριε Ποστήλε, εσείς. Σας ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Λάγκε. Ναι, νομίζω καλή ιδέα θα ήταν να πλουστεύσουμε κάπως τον πίνακα για τις εφαρμογές. Έχουμε εθελοντικού χαρακτήρα στοιχεία για τι τις και έχουμε τρεις κλίμακες ε, Euro 1, 2, 3. Καλή ιδέα θα ήταν οι δύο πρώτες φάσεις ε, να μπορέσουν να παγιωθούν, να χρησιμοποιούνται για να έχουμε περισσότερο χρόνο, περισσότερο περιθώριο στη βιομηχανία να αντιμετωπίσει προκλήσεις. Αυτό ταυτόχρονα θα έδινε κάποιες δυνατότητες και για την τελευταία, την ύστερη φάση, να δούμε πώς θα μπορούσαμε να επισπεύσουμε και τις ημερομηνίε Για τα μοτοποδήλατα είδαμε την, και την περίπτωση εκείνου του μοτοποδηλάτου που απέτυχε στις ε, δοκιμές ε, δίχρονου κινητήρα. Είχαμε άλλους κινητήρες που ανταποκρίθηκαν. Οι ε, εκπομπές ρήπων είναι πάρα πολύ υψηλέ όσον αφορά τους δίχρονους κινητήρες αυτά τα μοτοποδήλατα. Ευχαριστώ. Okay. Uh, Ευχαριστώ. Νομίζω θα μπορούσαμε να επανέλθουμε σε κάποια από αυτά τα στοιχεία υστερότερα. Αν δεν υπάρχουν τώρα άλλες ερωτήσεις, ας περάσουμε στη συνέχεια στον τελευταίο γύρο, στις τελευταίες παρουσιάσεις και θα έχουμε μετά ένα γύρο που και οι ομιλητές θα μπορέσουν να παρεμβούν. Για τον τελευταίο γύρο θα δούμε κάποια θέματα για την εφαρμογή, implementation των νέων Έχουμε τον κύριο Περλό που είναι υπεύθυνο ε, των ε, δημοσίων ε, αυτών σχέσεων και θεμάτων για τους ευρωπαϊκούς κατασκευαστές μοτοσυκλετών και θα μας δώσει κάποια στοιχεία σχετικά. Και ένα πράγμα, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Αντώνιο Περλό στην αρχή. Είχαμε μια ερώτηση του κυρίου Ρούιλε για το κόστος των συστημάτων ABS. Ίσως αυτό Ξέρω ότι έχετε κάποιες παρατηρήσεις που θέλετε να κάνετε. Σω θα μπορούσατε σε κάποια φάση να τοποθετηθείτε σε σχέση και με αυτό το θέμα, ε, σε σχέση με τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας. Έχετε τον λόγο κύριε Αντώνιο Πέρλο, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ που μας δίνετε την δυνατότητα να κάνουμε μια δήλωση σε αυτή τη δημόσια ακρόαση από πλευρά μα. Γίνεται μεγάλο λόγο για τι προκλήσει και τι πρέπει να κάνει η βιομηχανία. Γίνεται λόγο για ένα ασφαλέ περιβάλλον. Συχνά. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρω είναι πώς αυτές οι προκλήσεις αντιμετωπίζονται, μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα σε ένα χρονοδιάγραμμα, σε ένα χρονοπλαίσιο, κάποια στοιχεία σε σχέση με το γράφημα που μπορείτε να δείτε που συνδέει τους ε, κύριους παραγωγούς ε, που ε, παράγουν εξαρτήματα σε σχέση με αυτά τα οχήματα. 90% στην παραγωγή έχουμε ποσοστό, 80% της ευρωπαϊκής παραγωγής και κατασκευαστές που δεν είναι παραδοσιακά Ευρωπαίοι, Κάποιοι από αυτούς έχουν και βιομηχανεί και έδραση στην Ευρώπη. Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Όπως προανέφερα για τον κανονισμό, υποστηρίζουμε συνολικά τους στόχους για την στρατηγική Ευρώπη 2020. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υποστηρίζουμε τους τέσσερις ε, κύριους στόχους που κυρίω είναι απλούστευση, ασφάλεια, σεβασμός του περιβάλλοντος και νέες διοικητικές απαιτήσει ε, είναι μια πρόκληση για τους βιομηχανικούς κύκλους. Ε, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα εντάσσεται και μια μεγαλύτερη περιπλοκότητα όσον αφορά τα κράτη-μέλη που θα πρέπει να αδειοδοτούν και επίσης έχουμε τεχνικές προκλήσεις υπό το πρίσμα της παραγωγής αλλά και της διάθεσης στις αγορές γιατί θα πρέπει να πολλούνται στο τέλος τέλος αυτά τα οχήματα σε πελάτες. Ποιες είναι οι ε, προβλέψιμες επιπτώσεις για το κόστος, υψηλότερο κόστος ε, για, για μια δεκαετή περίοδο που καλύπτεται για παράδειγμα από τον κανονισμό Επίσης έχουμε σχεδιασμό, έρευνα, ανάπτυξη, σχετικές δαπάνες ως σκέλος που και αυτές λαμβάνονται υπόψη. Αυτές οι προκλήσεις σημαίνουν ότι το περιθώριο για το χρονοδιάγραμμα είναι θεμελιώδους σημασίας και για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις και για τον τομέα παραγωγής αλλά και για τους καταναλωτές. Επόμενο γράφημα. Γίνεται λόγος για διαφορετικές μορφές και τύπους οχημάτων στην ευρωπαϊκή αγορά. Πολύ συχνά συνδέουμε αυτό με μεγάλες μοτοσυκλέτες. Θα πρέπει να τονίσουμε όμως ότι πάνω από το ίμιση της αγοράς αποτελείται από σκούτερ και έχουμε και χαμηλής υποδύναμης ε, ε, μοτοποδήλατα που και αυτό είναι σημαντικό ε, στοιχείο στη διαφοροποίηση αυτή. Επόμενο γράφημα παρακαλώ. Δύο λόγια δεν είναι πολύ σαφές αυτό εδώ, αλλά δύο λόγια για το περιθώριο και το ε, χρονικό, τη χρονική δυνατότητα που θα έχουμε στη διάθεσή μας να δράσουμε κάποιες τοποθετήσεις ε, σε σχέση με τον μέσο κύκλο ζωής μιας μοτοσυκλέτας που μπορεί να είναι περίπου 10 χρόνια ανάλογα με τον τύπο. 3 3-4 χρόνια χωρίς ε, μεγάλες αλλαγές μετά μια ε, ε, ε, στην ημιπερίοδο κάποιες σημαντικές αλλαγές και αν δει κανείς την οικονομία κλίμακας που αναφέρθηκε προηγούμενα πρέπει να τονίσουμε το καλύτερο μοντέλο που πωλείται είναι στον αριθμό 20.000 μονάδων ετήσια για να δώσω ένα, μια μονάδα σύγκριση ε, για το πιο επιτυχέ αυτοκίνητο κάνουμε λόγο για πάνω από 500.000 μονάδε γιοταχή. Έτσι έχουμε περίπου ε, άλλε ε, που βρίσκονται, άλλα προϊόντα που βρίσκονται κάτω από 5.000 μονάδων ετήσια. Αυτό τι σημαίνει σε σχέση με την διαχείριση της δυνατότητας παραγωγής κατά μέσο όρο. Μπορούν να έχουν 30 διαφορετικού κινητήρε τέτοιου είδου προϊόντα. Αυτό περιπλέκει τα πράγματα. Υπάρχουν 20 έως 40 διαφορετικά μοντέλα, τύποι. Και γιατί συμβαίνει αυτό, διότι υπάρχουν ε, διαφορετικοί σκοποί και ε, ε, λόγοι χρήσης, καθώς επίσης και για τις απαιτήσεις των χρηστών. Δημιουργείται μεγάλος κατακαιρματισμός όσον αφορά μια οικονομία κλίμακας για αυτόν τον τομέα. Από την άλλη πλευρά έχουμε και ουσιαστικά τον χαρακτηριστικό σχεδιασμό ε, δυνατότητας παραγωγής. Ένα έτος ε, είναι ο χρόνος που χρειάζεται για την ανάπτυξη μιας τέτοιας, ε, ενός τέτοιου νέου προϊόντος. Μετά ακολουθούμε μια τετραετή περίοδο με ίσονο σημασία αλλαγές και μια επόμενη περίοδο που ακολουθεί μεγαλύτερων αλλαγών. Επόμενο γράφημα παρακαλώ. Εδώ έχουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μπορείτε να δείτε ουσιαστικά αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι μια ολόκληρη σειρά απαιτήσεων κάποιες από αυτές τις απαιτήσει ακολουθούν μια πολύ λογική προσέγγιση και δομή. Υπάρχουν διαφορετικές ημερομηνίες που προβλέπονται για τα διαφορετικά, τις ευρω, διαφορετικές ευρωφάσεις, Eurosteps και υποστηρίζουμε αυτές. Υπάρχουν ωστόσο και διαφοροποίησεις που γίνονται για νέου είδους αδειοδοτήσεις. Πράγμα πολύ σημαντικό, διότι η προσαρμογή σε σχέση με τις αδειοδοτήσεις συνεπάγεται ακόμα μεγαλύτερο έργο για μας. Αλλά δεν είναι αυτές όλες οι απαιτήσει που απαιτούνται. Όπως προαναφέρθηκε η απέτηση για το ABS υφίσταται αυτή τη στιγμή υφίσταται αυτό για όλα τα νέα οχήματα, για όλες τις νέες μοτοσυκλέτες από μια συγκεκριμένη ημερομηνία και πέρα και αυτό περαιτέρω περιπλέκει την παραγωγή τέτοιων προϊόντων. Ποια μπορεί να είναι η επίπτωση για τους παραγωγούς. Έχουμε πολύ στενό χρονικό περιθώριο για να προσαρμοστούμε. Αναφέρθηκε από τον κύριο Φαντεκάμπ σε αυτό. Δημιουργούνται καθυστερήσεις, υπάρχει ε, θέμα χρο, ε, χρονικής ε, καθυστέρησης και στο Συμβούλιο. Αλλά τα πράγματα δεν έχουν ε, προχωρήσει όπως αναμέναμε. Αν δεν προχωρήσουμε ταχύτερα δεν θα μπορέσουμε καν να ανταποκριθούμε στην απέτηση τη ημερομηνία του 2013 όπω προβλεπόταν την πρώτη πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επόμενο γράφημα. Ουσιαστικά αυτή είναι η περίληψη των αλλαγών που προτείνει η ΑΣΕΜ. Αυτός ο κύριος στόχος είναι να εξορθολογικευθεί το χρονοδιάγραμμα, να μπορέσουμε να θέσουμε σε δέσμες κάποιες απαιτήσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, μπορείτε να το δείτε σε αυτό το γράφημα. Ουσιαστικά προτείναμε να μεταθέσουμε την εφαρμογή του κανονισμού κατά ένα έτος, τουλάχιστον, τουλάχιστον, θέλω να το πω αυτό ξεκάθαρα. Είναι μια δυναμική διαδικασία. Μετεξελίσσονται τα πράγματα. Δεν υπάρχει καμιά εγγύηση. Δεν υπάρχουν εχέγγυα για την τελευταία δέσμη μέτρων. Όχι μόνο για αυτήν την απόφαση που βρίσκεται υπό τη διαδικασία συναπόφαση, αλλά και για την ολοκλήρωση. Η προβλεψιμότητα είναι σημαντική για να μπορέσει κανείς ε, στο σχεδιασμό να αναπτύξει ένα τέτοιο προϊόν. Άφησα στο άνω μέρος του γραφήματος ε, τον κύκλο ζωής που προανέφερα. Ήδη βρισκόμαστε στην κατάσταση που θα πρέπει να συμπυκνώνεται πάρα πολύ η φάση σωστής ε, ε, ορθολογικής ανάπτυξης και αν συμπυκνωθεί ακόμα περισσότερο θα είναι ανέφικτο να ανταποκριθούμε στις απαιτήσει ε, από πλευρά Η άλλη σημαντική πτυχή που υπάρχει εδώ είναι ουσιαστικά το ότι εφαρμόζεται η λογική ουσιαστικά Πρώτον, να εφαρμόζονται αυτές οι απαιτήσει σε όλες τις νέες αδειοδοτήσεις και για όλους τους νέους τύπους ε, ABS και OBD για να μπορούν οι αλλαγές σε μια φάση να μπορέσουν να εγκριθούν και να εφαρμοστούν. Είναι πολύ σημαντικό και για τους παραγωγούς αλλά και για τα κράτη-μέλη. Υπήρχαν αυξημένε ανησυχίες για τις περιπλοκές που θα μπορούσε να συνεπάγεται μια τέτοια ρύθμιση ενός τέτοιου κανονισμού. Καθώς επίσης και τις πληροφορίες για την ε, ε, συντήρηση και για, τις, ε, για τα συνεργεία και τις ε, ε, επισκευές που θα απαιτούνται. Όλα αυτά ως προϋποθέσεις είναι πολύ δύσκολο να ανταποκριθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε τέτοιο φόρτο εργασίας, ιδιαίτερα μέσα στο πλαίσιο των απαιτήσεων για τις μοτοσυκλέτες. Γι' αυτό λέμε θα πρέπει να μετακινηθεί το 2000 ε, από το 2017 να φτάσουμε ίσως το 2020 για κάποιες από αυτές τις απαιτήσει. Έτσι θα μπορέσει να μειωθεί η πίεση σε σχέση με τους ε, παραγωγούς και θα δοθεί μεγαλύτερη δυνατότητα. Θα υπάρξει περισσότερος χρόνος να μέσα σε ένα ορθολογικό πλαίσιο να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις και να ελέγξουμε και το κόστος, το οποίο είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Θα έχουμε ένα διαχειρίσιμο πλέον πλαίσιο όσον αφορά την δράση το, για τους παραγωγούς πολύ σημαντικό στοιχείο. Επόμενη τελευταία διαφάνεια παρακαλώ. Το προανέφερα αυτό. Αυτή θα ήταν η κατάσταση που θα απαιτεί σε μια ιδανική κανονική ομαλή κατάσταση της αγοράς. Καθώς γνωρίζετε έχει υποστεί σημαντικότατα πλήγματα από την κρίση η βιομηχανία. Χάσαμε 25% της αγοράς τα τελευταία, την τελευταία περίοδο και δεν υπάρχει κάποιο μήνυμα, κάποιο σημείο ανάκαμψης. Και να σας πω ότι η αυτοκινητοβιομηχανία κατά την ίδια περίοδο απόλυσε μόνο 6%. Απολέσαμε εμείς τις μοτοσυκλέτες πάνω από 4 φορές τετραπλάσιο ποσοστό ε, όσον αφορά την παραγωγή των μοτοσυκλετών. Και αυτό έχει τεράστια σημασία όσον αφορά τη μελλοντική προοπτική. Αυτή ήταν η τελευταία που διαφάνεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Uh, Mr. Bassett. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, θα σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δίνεται να σας παρουσιάσουμε τις παρατηρήσεις μας όσον αφορά την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε υπεύθυνοι για την παροχή υπηρεσιών και διανομή ανταλλακτικών μετά την πώληση και βεβαίως θέλουμε να αντιδράσουμε σε όλες τις κατηγορίες. Καταρχήν πρέπει να πω ότι μας αφορά να υπάρχει ανταγωνισμός, θεμητός ανταγωνισμός ε, σε όλες τις ε, κατηγορίες ε, και την παροχή υπηρεσιών. Καταρχήν να σας πω ότι με, για τις υπηρεσίες μετά την πώληση υπάρχουν 37.000 σημεία πώληση και παροχής υπηρεσιών στην Ευρώπη. 37.000 λοιπόν και 150.000 εργαζόμενοι. Πρόκειται για το 72% του όλου κύκλου εργασιών. Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι ότι ουσιαστικά μετά την πώληση υπάρχει μια ολόκληρη αλυσίδα φορέων παροχής υπηρεσιών για τα δίκυκλα μηχανοκίνητα και στην αρχή της αλυσίδας αυτής υπάρχει ο πολιτής, αυτός που παρέχει υπηρεσίες συντήρησης, επισκευές που παρέχονται σε όλη την αλυσίδα για όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος. Θα ήθελα εδώ να μοιραστώ μαζί σας κάποιες ιδέες όσον αφορά τον σύγχρονο τρόπο επισκευής, συντήρησης ε, μηχανοκίνητων ε, δίκυκλων οχημάτων. Τι γίνεται παραδείγματος χάρη σε ένα συνεργείο. Ο εντοπισμός του οχήματος διάγνωση, ε, εντοπισμός των προβλημάτων, σωστή ανάλυση του προβλήματος, εμπειρογνωμοσύνη, σύγχρονη, εντοπισμός των ανταλλακτικών που έχουν το πρόβλημα, σωστή αντικατάσταση των ανταλλακτικών, παραγγελία, επισκευή και στο τέλος βεβαίως θα πρέπει να ασχοληθεί κανείς με τα σύγχρονα τμήματα του οχήματος, το λογισμικό και την δυνατότητα να μπορέσει ο οδηγός να πάρει το όχημά του και να το οδηγήσει μετά την επισκευή. Χρειάζεται λοιπόν μία έγκαιρη και σύγχρονη διάγνωση, άρα πρόσβαση σε τεχνικές πληροφορίες και βεβαίως OBD συστήματα απαιτούν απαραίτητη τεχνική κατάρτιση και όλοι αυτοί οι οποίοι καθημερινά κάνουν τέτοιου είδους επισκευές και συντηρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν τα ανταλλακτικά και τα μηχανήματα όλων των τύπων. Η συντήρηση και η επισκευή θα πρέπει να βασίζεται σε όλες αυτές τις κατηγορίες, κατάρτιση, ανταλλακτικά, επισκευές και βεβαίως εργαλεία που να ανταποκρίνονται σε όλους τους τύπους και τις μάρκες. Εδώ βλέπετε που βρίσκεται η τεχνική πληροφορία, ποιες είναι οι πηγές, η πρόσβαση. Ο κατασκευαστής οχημάτων είναι αυτός ο οποίος έχει όλες τις τεχνικές πληροφορίες. Αριστερά βλέπετε την τακτική κανονική ενημέρωση, πληροφορία που χρειάζεται για την επισκευή και δεξιά βεβαίως θέματα συμβατότητας, ανταλλακτικών, τμήματων, μηχανημάτων. Τα ανταλλακτικά, τα μηχανήματα, ο εξοπλισμός για τη σωστή διάγνωση, ανάλυση και βεβαίως ανταλλακτικά και μηχανήματα και εργαλεία τα οποία ανταποκλίνονται σε όλους τους τύπους και τις μάρκες μηχανών και μοτοσυκλετών. Όλη αυτή η πληροφορία είναι απαραίτητη για να γίνει σωστή επισκευή. Όσον αφορά τα μακροοικονομικά στοιχεία, είναι πολύ σημαντική η πτυχή ασφάλειας και περιβαλλοντολογικής συμμόρφωσης και θα πρέπει να είμαστε στη θέση να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει η συμμόρφωση για όλη τη διάρκεια ζωής ε, του οχήματος και βεβαίως να διατηρήσουμε έναν θεμητό και αποτελεσματικό ανταγωνισμό σε όλες αυτές τις ε, προσφορές υπηρεσιών προς όφελος των καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως να υπάρχει συνοχή στην ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Μιλάμε σήμερα για τα πρότυπα Euro 5, Euro 6, ο εισηγητής αναφέρθηκε στις κατηγορίες οχημάτων λάμδα, τι και βεβαίως η συνοχή θα πρέπει να υπάρχει σε όλη την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και την σκοπιμότητα και το κατά πόσο είναι εφικτό αυτό το χρονοδιάγραμμα. Ιανουάριος του 2013 θεωρούμε ότι αυτό είναι πολύ εφικτό χρονοδιάγραμμα. Σήμερα πάνω από το 90% της ε, αγοράς ε, καλύπτεται από πολύ μεγάλους ε, οργανισμούς, μάρκες, κατασκευαστές όπως η Honda και Yamaha και άλλοι. Όλοι οι κατασκευαστές ήδη έχουν τις τους, ε, τα δικά τους δίκτυα παροχής υπηρεσιών και βεβαίως σήμερα πρέπει να πούμε ότι η κρίση πλήττει τον τομέα, πλήττει ιδιαίτερα τις ε, παροχές υπηρεσιών μετά την πώληση. Ζητάμε λοιπόν σήμερα κοινά πρότυπα, αλλά βεβαίως αυτό δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Και βεβαίως η πληροφορία που ζητείτε για την έγκριση τύπου είναι μια πληροφορία που βεβαίως μπορεί να ζητηθεί, να δοθεί και μετά υπάρχει ένα εξάμεινο έτσι ώστε να υπάρξει η συμμόρφωση. Όσον αφορά τα πρότυπα Euro 5 και Euro 6 λατινικό, χρειάζονται σαφείς βελτιώσεις σε σχέση με το πρώτο κείμενο της Επιτροπής, ε, η οποία το 2000 επέβαλε κάποια πρότυπα, που βεβαίως είχαν εμπνευστεί από την ε, αυτοκινητοβιομηχανία. Υπάρχει σήμερα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης, σε αυτό νομίζω συμφωνούμε όλοι. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να σας παρουσιάσω αυτή την τελευταία διαφάνεια. Το μόνο που τελικά ζητάμε είναι να μπορέσουν όλοι οι φορείς παροχής υπηρεσιών να συνεχίσουν να εργάζονται σε ένα κλίμα, μια ατμόσφαιρα θεμητού αποτελεσματικού ανταγωνισμού και πιστεύουμε ότι μέχρι το 2016-2020 θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες και δεν νομίζω ότι θα πρέπει εγώ να επανέλθω σε θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ. Μέσα σε 8 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα ξεπετάξατε τα επιχειρήματά σας. Δεν χρειάζονται περισσότερα λόγια. Αυτά που θέλετε να πείτε τα είπατε και μας βοήθησαν πολύ. Έχουμε χρόνο για ένα γύρο ερωτήσεων Τώρα, αν θέλετε να θέσετε ευρύτερα θέματα, δεν έχουμε το χρόνο. Ε, δεν μιλήσατε για το κόστος του ABC, του ABS, συγγνώμη, της κυρίας Ρούλε. Δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε τώρα ή να περιμένετε πρώτα και τις άλλες ερωτήσεις να απαντήσετε μαζί. Για τον κύριο Έχουμε λίγο χρόνο από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούμε να του δώσουμε λίγο χρόνο για να κάνει μια παρέμβαση. Πέντε λεφτά θα του δώσουμε πριν από το τέλο τη ακρόασή μα, αν συμφωνεί. Τώρα θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους και θα ήθελα να δώσω και το λόγο στον κύριο Βάντεν Κάμπ για να συνοψίσει στο τέλος. Ο κύριος Λάγκ, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Πράγματι πρόεδρε, πιστεύω ότι πρέπει κάποια σημεία να τα δούμε ακριβώς σε βάθος, σε λεπτομέρειες. Στον προηγούμενο γύρο κατέστη φέσο ότι παράλληλα στο θέμα των οριακών τιμών υπάρχει και το θέμα της αηφορίας και του ε, κύκλου ζωής ε, και της διάρκειας ζωής, πράγμα το οποίο έχει αποφασιστική σημασία και σε κάποια δέκατα ή ε, εκατοστά της ορια, των οριακών τιμών δεν θα έδινα τέτοια μεγάλη σπουδαιότητα όπως στον κύκλο ζωής όπου για κάποια οχήματα μετά από κάποια χιλιόμετρα δεν αντέχουν στις προδιαγραφές και δεν τα βγάζουν πέρα. Είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και τίθεται το θέμα πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε μακρό κύκλο ζωή. Και εδώ φτάνουμε πραγματικά στο OBD, στο σύστημα OBD, on board ε, εξοπλισμού και τη εποπτείας της αγοράς. Και θα μπορούσα να φανταστώ πώς πιο σαφείς κανόνες και κανονισμοί θα έπρεπε να εξευρεθούν για να λειτουργήσουν σωστότερα τα πράγματα ώστε αυτή η απέτηση της μακρότερης ζωής ε, ενός προϊόντος να μπορεί να ε, διασφαλιστεί. Και υπό αυτό το πρίσμα, κύριε Πρόεδρε, υπό το πρίσμα του εισηγητή πρέπει να προβληματιστεί κανείς κατά πόσον η επιτροπολογία μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί για να ρυθμίζει προβλήματα. Στον τομέα του ιόταχή και της νομοθεσίας έχουμε το Euro 5 και το Euro 6 αλλά και στην νομοθεσία για τα φορτηγά έχουμε παρόμοιες κλίμακες δίνεται μεγάλο πλαίσιο στην επιτροπολογία μεγάλη δυνατότητα παρέμβασης πράγμα το οποίο όσον αφορά τις διαδικασίες πρέπει να ληφθεί υπόψη όσον αφορά τον χρονορίζοντα και για τις εκπομπές ρήπων υπήρξαν τριβές και προβλήματα. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι στην κοινοβουλευτική διαδικασία τέτοιου είδους προδιαγραφές και ε, μηχανισμοί εποπτείας πρέπει να διασφαλίζονται και να κατοχυρώνονται. Εδώ κοινοβουλευτικά πρέπει να δούμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε και να περιορίσουμε τη διαδικασία της επιτροπολογίας, να μην έχει τέτοιο εύρος. Τρίτο, βρήκα η παρουσίαση σε σχέση με τους παραγωγούς ανταλλακτικών και εξαρτημάτων πιστική. Με το Euro 4 για τα ΙΟΤΑΧΗ έχουμε απαιτήσει που τίθενται για την προσπελασιμότητα των τεχνικών, τεχνολογικών πληροφοριών και στοιχείων και πρέπει αυτό να το προωθήσουμε και να το προσαρμόσουμε, διότι οι αρχές είναι οι ίδιες, αλλά οι τεχνολογικές δυνατότητες έχουν αλλάξει και το τι είναι δυνατό να γίνει έχει αλλάξει. Πρέπει να διασφαλίσουμε οι τεχνολογικές αξίες και ε, ε, τα τεχνολογικά στοιχεία και δεδομένα να έχουν διάθεση στους πολίτες να μπορούν ε, σε ανεξάρτητα συνεργεία να επισκευάζουν τα οχήματά τους οι πελάτες. Η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές πρέπει να βελτιωθεί όσον αφορά τον χρονορίζοντα και τα χρονικά περιθώρια, Αντώνιο, πρέπει να προβληματιστούμε και να δούμε αν μπορούμε να εναρμονίσουμε τα πράγματα κάπως. Σημαντικό όμως θα είναι να προσδιορίσουμε ποια είναι τα στοιχεία κλειδιά, τα κυριότερα σημεία. Και θα ήθελα να συζητήσουμε σε αυτό το χρονορίζοντα να δούμε αν αυτό θα είναι η πορεία που θα ακολουθήσουμε και με ποιο τρόπο. Ευχαριστώ. If Θυμάμαι καλά για τον εναρμονισμό για τον τρόπο της παραγωγής και παρουσίασης στοιχείων ήταν κέρια σημασία στοιχείο ε, όσον αφορά για ή επιβατικά αυτοκίνητα. Θα πρέπει να το δούμε αυτό κυρία, ε, και από πλευρά της κυρία Ρούλε είχε τεθεί. Κυρία Ρούλε, έχετε κάποιες αρετήσεις, εσείς σχόλια. Η κυρία Ρούλε Και εγώ θέλω να επιμείνω περισσότερο σε αυτό, γιατί και εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις μεταξύ του δεύτερου γύρου και του τρίτου γύρου. Αν κατάλαβα καλά τα όσα είπε ο δεύτερος γύρος και οι δύο επαΐοντες ξεκάθαρα σχετικά είπαν ότι υπάρχει η δυνατότητα να απαιτούνται υψηλότερες προδιαγραφές. Είναι ε, αυτό μια δυνατότητα. Έτσι λοιπόν όσον αφορά τις τεχνικές δυνατότητες ε, διανοίγονται νέες δυνατότητες. Και αν κατάλαβα καλά και ερμηνεύω τον δεύτερο γύρο σωστά, υπήρχε η επιθυμία να εναρμονιστούν κάποιες ε, ε, διαδικασίες, αλλά να μην μετατεθούν οι χρονοορίζοντες. Στον τρίτο γύρο ακούσαμε μετάθεση ημερομηνιών. Θέλω να ε, απευθύνω την ερώτηση στους παραγωγούς ανταλλακτικών και εξαρτημάτων τι θα γίνει. Με αυτή την ε, ε, μετάθεση ημερομηνία είναι η καλύτερη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε την κρίση και τις προκλήσεις. Να θυμόμαστε ότι δεν έχουμε μόνο παραγωγούς στην Ευρώπη αλλά και στην Ινδία και στην Κίνα όπου η επιβάρυνση του περιβάλλοντος μέσω μοτοσυκλετών έχει φτάσει υψηλότατες τιμές και έχει, επιδεινώσει το, έχει επιδεινωθεί η κατάσταση του περιβάλλοντος. Να δούμε μήπως αποκομίσουν αυτοί προτερήματα, πλεονεκτήματα όσον αφορά τον ανταγωνισμό και στρεβ στρεβλώνεται η ανταγωνιστική μας θέση. Να τα δούμε αυτά, να συγχωνεύσουμε ίσως κάποιες διαδικασίες, αλλά μην μεταθέσουμε. Κύριος Ρεπότ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ο κύριος Ρέπο, ευχαριστώ τους επαΐοντες και οι επαΐοντες προφανώς πάρα πολλά έδωσαν ω στοιχεία, τεχνολογικής, τεχνικής μορφής στοιχεία. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στην τελευταία παρέμβαση που έγινε. Ποιος κίνδυνος υφίσταται, θεωρείτε εσείς, τι θα λέγατε, ποιος είναι ο κίνδυνος όταν έχουμε την προπαρασκευή, για παράδειγμα, της πέμπτης κλίμακας ε, Euro 5, πώς μπορεί κανείς να μεριμνήσει και να διασφαλίσει ώστε η περίοδος αυτή να, να τηρηθεί χρονικά. Και τι γίνεται με την ανταγωνιστικότητα, με τις λύσεις για τον ανταγωνιστικό όσον αφορά την Ευρώπη, όσον αφορά τις δυνατότητες διάθεσης στην αγορά. Ευχαριστώ. Uh, Το είναι θέμα βιομηχανικής πολιτικής. Ως κοιόδης να κάνω και εγώ κάποια σχόλια. Θέλω να επανέλθω στις τελευταίες δύο παρουσιάσεις για την επισκευή και τη συντήρηση. Ο κύριος Μπασέ ε, είπε κάτι ενδιαφέρον είπε για τις τέσσερις βασικές αρχές της μοντέρνας επισκευής. Κατάρτιση και πληροφορία ε, για τις επισκευές και την συντήρηση. Οι κατασκευαστές, κατά τη γνώμη σας, πώς θα μπορέσουν να ελέγξουν ότι τα συνεργεία στα οποία δίνουν τις ε, πληροφορίες ε, καταρτίζονται σωστά, έχουν τα εργαλεία και έχουν και το, τη δυνατότητα να διαδώσουν αυτές τις πληροφορίες. Ε, δεύτερη ερώτηση προς τον κύριο Περλό. Αν σας ικανοποιώ ως ε, κατασκευαστής ότι έχω δηλαδή την απαραίτητη κατάρτιση, τα απαραίτητα εργαλεία και τις πληροφορίες, τότε θεωρούμε εγκεκριμένο συνεργείο. Μπορείτε να με θεωρήσετε να με διορίσετε ως εγκεκριμένο συνεργείο, ας πούμε. Κάτι που θέλω να απευθύνω κυρίως στον κύριο Περλό. Δεν νομίζω ότι απαντήσατε ένα σημαντικό ερώτημα του κυρίου Λάγκετ και της κυρίας Ρούλε για το αν χρειαζόμαστε αυτά τα euro. Χρειαζόμαστε αυτό το euro 4, 5 και 6 και να το εφαρμόσουμε σε μια τόσο σύντομη χρονική περίοδο. Ε, με βάση τις παρουσιάσεις που έγιναν, που είναι πολύ πιστικές, προκύπτει ότι τα οχήματα ε, ήδη έχουν επιδόσεις που ξεπερνάνε το Euro 4, ήδη σήμερα. Θα κάναμε εξοικονόμηση χρόνου, αν λέγαμε στην ε, Κομισιόν ότι δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Ίσως θα πρέπει να δούμε λοιπόν αυτό το θέμα της πρότασης σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, Πρόεδρε, μία ερώτηση, μία ερώτηση μόνο. Και στον, προς τον κύριο Λουκ, ε, όσον αφορά την ε, πολιτική κατά του τάμπερινγκ. Στην παρουσίαση σας είπατε ότι το πείραγμα μηχανών είναι μεγάλη απειλή για το περιβάλλον και απειλή και για την ασφάλεια ιδιαίτερα όσον αφορά εκείνους που έχουν μοτοποδήλατα, σκούτερ, όλοι είμαστε κάποτε νέοι και όλοι θυμόμαστε τι γινότανε, πειράζαμε τα δίκυκλά μας, τους κινητήρες τους. Τι κάνετε εσείς στη Γαλλία για να αντιμετωπιστεί το πείραμα εντός εισαγωγικών κινητήρων. Δεν θέλω να έχουμε μια αποκλειστική εμβάθυνση σε αυτό, αλλά θέλω να ξέρω τι γίνεται με τα μέτρα αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Έχουμε 10 λεπτά όλα όλα και θέλω να δώσω και λίγο χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι διερμηνείς κάποια στιγμή πρέπει να φύγουν λοιπόν. Τι θα κάνω λοιπόν. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπασέτ και στον κύριο Περιλό. Θα τους δώσω δύο λεφτά στον καθένα. Μετά θα δώσω το λόγο ε, για ένα λεπτό σε οποιοδήποτε από τους άλλους ε, βασικούς ε, φιλοξενούμενους. Και δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κύριος Μπάστερ πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο καλύτερα μπορώ. Μία ερώτηση. Ε, πώς γίνεται κανείς εγκεκριμένο συνεργείο. Πολλοί από τα, πολλά από τα συνεργεία δεν θέλουν να είναι τμήμα αυτού του κυκλώματος, ε, εγκεκριμένα συνεργεία. Είναι θέμα επιλογής των κατασκευαστών. Μερικές φορές δεν θέλουν ε, ε, ένα συνεργείο να επιδιορθώνει ε, μοτοσυκλέτε πολλών διαφορετικών προελεύσεων. Όπως σα είπα, το κύκλωμα αυτό είναι πραγματικό κύκλωμα μετά την πώληση. Χρειαζόμαστε τεχνικές πληροφορίες ε, για τα ε, εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι ανεξάρτητη, τα ανεξάρτητα συνεργεία που έχουν την ικανότητα γιατί έχουν τις πληροφορίες, έχουν την κατάρτιση, πώς θα, ότι θα τη χρησιμοποιήσουν σωστά. Ε, είναι θέμα ευθύνης. πρέπει κανείς να συμπεριφερθεί σωστά, να χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο αυτά που έχει, ε, να συντηρεί σωστά τα οχήματα. Πρέπει να γίνει σωστή κατάρτιση και είναι και θέμα και των οργανώσεων να εξηγήσουν ε, και να διαδώσουν τις πληροφορίες ότι χρειάζονται όλα αυτά τα πράγματα για να γίνει σωστή συντήρηση. Ε, το κάναμε μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής λειτουργούσαμε σωστά. Τώρα που έχουμε αυτό το τεχνολογικό, κάνει αυτό το τεχνολογικό άλμα, γιατί να αλλάξουμε. Ίσα ίσα θα πρέπει να συνεχίσουμε και καλύτερα μάλιστα. Αυτά ευχαριστώ. Δύο λεφτά, μέσα στην ώρα σας. Μπράβο. Και εγώ με χαρά θα κάνω το ίδιο. Υπάρχουν πολλέ ερωτήσει. Να ξεκινήσουμε την ερώτηση τη κυρία Τρούιλε για την, από ό,τι φαίνεται, αντίφαση σε σχέση με τους δύο γύρους ε, μεταξύ ASEM και ACC. Αυτό που πολύ σαφώς ε, εντοπίστηκε από πλευράς του κ. Μπόσελ σε σχέση με τις μετρήσεις ε, που έγιναν χωρίς απαιτήσει κύκλου ζωής και αυτό έχει τεράστια διαφορά που δημιουργείται. Το να ανταποκριθεί κανείς ε, στο κύκλο ζωής και στι δοκιμασίε θα έπρεπε να προσαρμοστούν οι παραγωγοί σε 50% υπό το πλαίσιο των, νόμιμων, ε, των νομικών αυτών απαιτήσεων για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Είναι μια πολύ σοβαρή τεχνολογική μορφής πρόκληση αυτό. Και έτσι αυτό υποθέτω μπορεί να απαντήσει και στο θέμα των τριών φάσεων. Χρειαζόμαστε πραγματικά αυτέ τι τρει φάσει. Αν σκεφτούμε και λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη να εκπέμπουν λιγότερους ρήπους, μικρότερους ρήπους ε, οι κινητήρες των δίκυκλων και πρέπει να υποβληθεί και αντίστοιχη πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την κατεύθυνση. Σημαντικό είναι, λόγω της καθυστέρησης ε, που υπάρχει, ότι δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα ε, σε ένα καθεστώς πίεσης η δυνατότητα προσαρμογής αυτών των κινητήρων κάποιοι πρέπει να προσαρμοστούν ή να περιοριστούν στη διαδικασία επιτροπολογίας ε, και άλλοι όχι. Οι τρεις φάσεις αυτό το οποίο προβλέπουν, οι δύο φάσεις, οι δύο φάσεις προβλέπουν μια ε, κατά 25% κάθε μία μείωση των εκπομπών ρήπων. Πρώτον. Δεύτερον, πιστεύουμε ότι αυτό ε, δίνει τη δυνατότητα μιας ομαλής προσαρμογής στις περιβαλλοντικές προδιαγραφές, λαμβάνοντας υπόψη και την ε, κατάσταση έκθυλης κρίσης στην οποία βρισκόμαστε. Τώρα και για το κόστος του ABS στα δίκυκλα που αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο. Πολύ σημαντικό θέμα και πρέπει να απαντηθεί αυτό. Υπάρχουν πληροφορίες που δίνονται στο Ευρωκοινοβούλιο που κάνουν λόγο για το κόστος για τον καταναλωτή καταναλωτή περίπου 100 ευρώ. Θα επιθυμούσαμε και εμείς να συνέβαινε αυτό, αλλά πληροφορία προς εμάς. Ο κόστος, ε, το κόστος για τους παραγωγούς σήμερα, για το hardware, hardware για να ενταχθεί ως η, ο εξοπλισμός ABS σε μια μοτοσυκλέτα είναι 250 ευρώ και πάνω. Λάβετε υπόψη και την προσαρμογή του συστήματος και δεδομένης της πολύ μεγάλης ποικιλία που υπάρχει όσον αφορά κινητήρες, αυτή η προσαρμογή είναι πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι για κινητήρες ε, γιοταχή. Απαιτεί πολύ μεγαλύτερο fine tuning, πολύ μεγαλύτερη λεπτή προσαρμογή σε λεπτομέρειες ε, και ε, στην λειτουργία του κινητήρα. Και αυτό συνεπάγεται κόστος. Αναφέρθηκε ότι η διείσδυση στην αγορά είναι σχετικά χαμηλή. Δεν θέλω να το διορθώσω αυτό. Τώρα βρισκόμαστε στο περίπου 50% των οχημάτων με προηγμένα συστήματα τροχοπέδησης. Και ο μεγαλύτερος κυλινδρισμός, ο μεγαλύτερο κυβισμός έχει ABS. Αυτό περίπου 35% σε σχέση με τις πωλήσει. Οι οικονομίες κλίμακος που θα μπορούσαν να επιτευχθούν έχουν ήδη σε κάποιο ποσοστό επιτευχθεί. Φτάνοντας τώρα σε κόστος 100 ή κάτω των 100 ευρώ για τον καταναλωτή δεν είναι αξιόπιστη πληροφορία για μας. Στρεφόμενος προς τις άλλες ερωτήσεις και θέματα. Το θέμα, συγγνώμη, έχω μακρηγορήσει υπερβολικά. Λοιπόν, επαρκούμε σε αυτά. Ευχαριστώ. Ποιος άλλος θα ήθελε να πάρει το λόγο, ναι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα κι εγώ. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Περλό. Τα είπα κι εγώ ότι τα στοιχεία αυτά δεν έχουν διάρκεια. Εγώ έβγαλα κάποιες από τις διαφάνειες της παρουσίασής μου για να μην ξεπεράσω το χρόνο που είχα. Υπάρχουν όμως δημόσιες πληροφορίες από τον Williams για την διάρκεια αυτών των στοιχείων και για την μη διάρκεια κάποιων άλλων στοιχείων. Θα ήθελα να το πω αυτό και σε σχέση με την αντικατάσταση κάποιων ε, ανταλλακτικών, κάποιων μερών και αυτό θα πρέπει να ειδωθεί στη διάρκεια του χρόνου. Θα προσπαθήσω και εγώ πολύ σύντομα να μιλήσω για την παρέμβαση στα ελαφρά οχήματα. Εγώ μιλούσα για τα μοτοποδήλατα, αλλά υπάρχουν βεβαίως και τα σκούτερ, υπάρχουν και οι μοτοσυκλέτες. Η επίπτωση αυτής της παρέμβασης για τη βελτίωση των επιδόσεων ένα από τα αποτελέσματα αυτών των παρεμβάσεων είναι ο θόρυβος ε, των εξατμίσεων. Και ξέρετε πολύ καλά ότι οι αστυνομικοί παρεμβαίνουν κάθε φορά που υπάρχουν δυνατότητες πάνω από το 50% των ε, ελαφρών οχημάτων, των μοτοσυκλετών, έχουν υποστεί τέτοιες ε, παρεμβάσεις για βελτίωση επιδόσεων. Ήταν 60% παλιότερα αυτό το ποσοστό. Για τα δίχρονα, τους δίχρονους κινητήρες είναι πιο εύκολη η Ξέρετε ότι για τους κινητήρες των μοτοποδηλάτων με ηλεκτρονικό ψεκασμό είναι πιο δύσκολη η παρέμβαση από ότι σε κινητήρες ψεκασμού καυσέριου. Για τα δίχρονα δηλαδή ε, μοτοποδήλατα υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβασης και τροποποίησης. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τις διαφάνειες που μας παρουσιάσετε και οποιοδήποτε θέλει θα τις βάλουμε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Τον ευχαριστώ που ήταν παρόν σήμερα. Δεν έχετε βέβαια πολύ χρόνο στη διάθεσή σας αλλά μπορείτε ενδεχομένως να σχολιάσετε κάποια από τα σημαντικά που ακούσαμε και τέλος θα δώσω το λόγο στον εισηγητή για να κάνει και εκείνος κάποιες παρατηρήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Ήρθαμε να ακούσουμε σήμερα και ακούσαμε και μάθαμε πολλά. Ελπίζω να μπορέσουμε και εμείς να συμμετάσχουμε στη συζήτηση αυτή κάποια στιγμή με επικοδομητικό τρόπο. Θα ήθελα να απαντήσω σε τέσσερις ερωτήσεις. Το κόστος ABS, ασφάλεια, εκπομπές και χρονοδιάγραμμα. Το κόστος του ABS. Βεβαίως είναι πάρα πολύ σωστή η ανησυχία. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία, αξιόπιστα στοιχεία όσον αφορά το κόστος του ABS για όλη την γκάμα των προϊόντων. Το κόστος λοιπόν του ABS υπολογίζεται εδώ με ένα μέσο, αν θέλετε, τρόπο. Αυτό όμως που σήμερα μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει μια αναλογία 3 προς 1 κόστος και αποτέλεσμα. Αλλά επαναλαμβάνω, πρόκειται για μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα πρέπει να εξετάσουμε. Τώρα, ασφάλεια σε σχέση με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Βεβαίως και είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της ανθρώπινης συμπεριφοράς, του συμπεριφοράς του οδηγού. Και βεβαίως οι επιπτώσεις μιας διαφορετικής συμπεριφοράς μπορεί να είναι πολύ θετικές όσον αφορά την οδική ασφάλεια. Η αποφυγή ατυχημάτων όμως δεν είναι πάντα δυνατή. Όποια και να είναι η συμπεριφορά του οδηγού, πολλές φορές ένα ατύχημα είναι αναπόφευκτο. Τρίτο, εκπομπές. Υπάρχει ένα πολύ παράδοξο στοιχείο όσον αφορά τις εκπομπές σωματιδίων και αυτό είναι κάτι που δεν θα πρέπει να το αγνοήσουμε. Ο καλύτερος τρόπος να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό είναι να δούμε πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε την πηγή ε, των σωματιδίων, δηλαδή τους υδρογονάνθρακες και να δούμε πώς μπορούμε να τα περιορίσουμε από την πηγή. Δεύτερον, το χρονοδιάγραμμα, η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου που έχει καθυστερήσει συνεχίζει να ε, εργάζεται και να επεξεργάζεται τις προτάσεις αυτές. Σας υπόσχομαι ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί, θα επιταχυνθεί και ελπίζω με πολύ επικοδομητικό τρόπο να μπορέσουμε να υποβάλουμε στο Κοινοβούλιο τις ε, προτάσεις. Εγώ άκουσα πολύ προσεκτικά ποιε είναι οι ανησυχίες. Δεύτερον, το θέμα του χρονοδιαγράμματος για την επιτροπολογία. Βεβαίως, και ξέρουμε ότι θα πρέπει να προετοιμαστεί η διαδικασία της Επιτροπολογίας, αλλά θα πρέπει επίσης εσείς να ξέρετε ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής θέλουν να μπορέσουν να δεσμευθούν επί του χρονοδιαγράμματος έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της Επιτροπολογίας και να είναι έτοιμοι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ που μας ακούσατε. Θα ήθελα να εξηγήσω για άλλη μια φορά ότι η επιτροπολογία, που είναι μια λέξη γνωστή εδώ στις Βρυξέλλες, σημαίνει ότι σε κάποιους τομείς όπου η νομοθεσία, οι κανονισμοί δεν είναι επαρκής και χρειάζεται ενημέρωση και ανανέωση και μεταρρύθμιση, υπάρχουν εμπειρογνώμονες οι οποίοι εξετάζουν τις ε, τροποποιείς αυτές για να διαπιστώσουν ότι δεν ξεπερνούν τις αρχικές προθέσεις ε, του νομοδέστη. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή, στον κύριο Βάντεγκαπ, ευχαριστώντα τον για την διοργάνωση αυτής της ακρόασης. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Στις 7 θα πρέπει να είμαι σε ένα δείπνο που οργανώνει Άσεμ. Δηλαδή, εδώ στις Βρυξέλλες, περίπου 30 λεπτά για να πάμε μέχρι εκεί. Καταλαβαίνετε ότι προσβλέπω σε αυτό το πολύ ευχάριστο δείπνο. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την γραμματεία, τον κύριο Ντεφρίς, τους συνεργάτες μου, τους βοηθούς μου, που μπόρεσαν να οργανώσουν εδώ αυτήν την ακρόαση αλλά και το δείπνο και βεβαίως συγκεντρώσαμε όλους τους μοτοσυκλετιστές εδώ χάρη στην εξαιρετική διοργάνωση αυτής της ακρόασης. Ακούσατε τα εισαγωγικά μου σχόλια, θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε αυτές τις προτάσεις και σε λίγες εβδομάδες θα υποβάλουμε το σχέδιο έκθεσης και βεβαίως σας περιμένω Περιμένω να υποβάλλετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Ένα σημαντικό ερώτημα του Μπέντ Λάγκε. Τι θα πρέπει να αφήσουμε στην Επιτροπολογία. Εγώ απαντώ πολλά, γιατί είναι τεχνικά τα θέματα και για έναν πολιτικό σαν και εμένα το θέμα είναι εξαιρετικά τεχνικό. Θα δούμε όμως, θα δούμε αν εμείς σαν πολιτικοί αντιμετωπίσαμε σωστά τα θέματα των κανονισμών που είναι δικά μας θέματα. Θα δούμε όμως τι είναι οι αρμοδιότητες των πολιτικών και τι είναι αυτά που θα αφήσουμε στην Επιτροπολογία. Σας ευχαριστώ πολύ. Well, thank you very much indeed. Um, thank you all very much. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ όλους σας για τη συμμετοχή. Ευχαριστώ όλους που μας παρακολουθούν στο διαδίκτυο όσοι είναι αυτοί. Προσβλέπουμε στο να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας αυτή μαζί σας στους επόμενους ε, μήνες. Ε, σας ευχόμαστε καλό βράδυ για όλους. Για τα μέλη της Κοινοβουλικής Επιτροπής θα συνέρχομαι και πάλι την Δευτέρα 11 Απριλίου στις 3 το απόγευμα 15.00 για την επόμενη συνεδρίασή μας. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.